Καλό μεσημέρι, συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Έχετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης μπροστά σας. Γνωρίζετε, υποθέτω, πως ε, τελειώνει η ενδιάμεση προεδρία μου, η προσωρινή προεδρία μου. Το... Η ομάδα των φιλελευθέρων ε, θα προτείνει έναν υποψήφιο και προτείνω να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη για να ξεκινήσουν οι εργασίες Επιτροπής μας αμέσως με την Προεδρία του Νέου Πρόεδρου πρέπει να γίνουν τα πράγματα επισήμω. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούν κάποιες, ε, κάποιοι κανόνες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να διαπιστώσουμε αν υπάρχει απαρτία των μελών το οποίο σημαίνει αν είναι παρόντες ε, το 1 τέταρτο των 29 μελών, δηλαδή αν υπάρχουν 8 συνάδελφοι, νομίζω πως υπάρχουν παραπάνω από 8 συνάδελφοι, οπότε έχουμε απαρτία και άρα μπορώ να ανακοινώσω την υποψηφιότητα ενός ε, νέου υποψηφίου Προέδρου. Η ομάδα των φιλελευθέρων προτείνει τον Γιάννη Μιλντερ που κάθεται εκεί στη δεύτερη σειρά. Ξέρετε πως μια υποψηφιότητα μπορεί να υποβληθεί από μια πολιτική ομάδα ή από έναν αριθμό βουλευτών. Αυτή τη φορά έγινε από την πολιτική ομάδα των φιλελευθέρων και δημοκρατών δηλαδή. πρέπει να ρωτήσω τον Γιάνν Μιλντερ εάν ε, αποδέχεται αυτή την πρόταση. Ναι, κύριε Πρόεδρε, βεβαίω. Καλώς, τότε πρέπει να ανακοινώσω πως ε, η γραμματεία εξέτασε αν εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις ο κύριος Μουλτερ και όσον αφορά και την δήλωση οικονομικών συμφερόντων έχουν δημοσιευτεί τα οικονομικά συμφέροντα του κυρίου Μιούλντερ στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, οπότε τα πράγματα φαίνεται πως είναι εντάξει. Οπότε θεωρώ πως είναι έγκυρη η υποψηφιότητα και αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να ρωτήσω είναι εάν υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι για την Προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού κανένας άλλος, οπότε ο κύριος Μιλντερ είναι ο μόνος υποψήφιος και εκτός εάν το 1 έκτο των μελών είναι κατά της υποψηφιότητας, κάτι το οποίο δεν βλέπω, νομίζω πως μπορούμε να εκλέξουμε ως νέο πρόεδρο διαβοής τον κύριο Μιλντερ. Εκτός εάν υπάρχει κάποιος αριθμός μελών. Eh, Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μίλντερ να καταλάβει τη θέση μου εδώ πέρα. Πρέπει να πω κύριοι συνάδελφοι και κύριοι συνάδελφοι πως ε, θα ήθελα, μια που βρίσκομαι ακόμα στο Δήμο, να πω πως χαίρομαι ιδιαίτερα για την εκλογή του κυρίου Μίλντερ. Μπορεί να μην το ξέρετε πως ε, ο Γιάνν βεβαίως είναι μέλος ε, εδώ και καιρό της ε, Επιτροπής μας και είναι ο πρεσβύτερος στην Επιτροπή, όχι πιο ηλικιωμένος, είναι ο συνάδελφος ο οποίος είναι, ήταν μέλος από το 1994 μέχρι το 2009, 15 χρόνια χωρίς διακοπή, ως ε, μέλος των ε, φιλελευθέρων, ε, έλαβε μέρος σε όλες τις συζητήσεις, στην πτώση Επιτροπής Σαντέρ μεταξύ άλλων, στην απάτη Τράνζιτ. Το 2009 δεν επανεξελέγει, αλλά επανήλθε τώρα και είναι πρόεδρος της Επιτροπής μας. Συγχαρητήρια Γιάννη. Ο κύριος Γκάιερ επίσης ζητάει το λόγο. Ήθελα μόνο να σου ευχηθώ συγχαρητήρια και καλή επιτυχία αγαπητέ Γιάν, εξ ονόματος της δικής μου πολιτικής ομάδας, αλλά θα ήθελα να πω ότι πάντως τα έκανε θαυμάσια και ε, ε, ε, πρότεινες εκπροσώπησης τον δικό μας εκπρόσωπο της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων των ε, συναδέλφων ως ε, κατά τη διάρκεια της θητείας σου ως προεδρέμων αυτής της Επιτροπής. <clears throat> Uh, για μια ακόμη φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την εκλογή μου στη συγκεκριμένη θέση. Σκοπεύω και ελπίζω να είμαι δίκαιος προς όλους, να μπορέσετε πάντα να εκφραστείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε μια ευαίσθητη επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης και πάρα πολλές αρμοδιότητες και έχει υποτιμηθεί ο ρόλος του σε σχέση με τα δημοσιονομικά της Ευρώπης εδώ και πολύ καιρό. Δεν ήμουν προετοιμασμένος για να γίνω πρόεδρος αυτής εδώ της Επιτροπής και γι' αυτό θα πρέπει να αποχωρήσω ήδη στις 5 σήμερα το απόγευμα γιατί η πατρίδα με καλεί. Αλλά με τον εξαιρετικό μου προκάτοχο εδώ θα με αντικαταστήσει επάξια γύρω στις 5. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και τον κύριο Στάες για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο προείδρευσε κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεταβατικής περίοδου. Μπορούμε να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη λοιπόν. Θα πρέπει καταρχάς να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Έχετε λάβει όλη την ημερήσια διάταξη. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Όχι, οπότε σε αυτή την περίπτωση υποθέτω ότι γίνεται δεκτή. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν στο σημείο 3. απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2009. Ποιος έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είχα παρακαλέσει πριν ε, περάσουμε σε κάποιες σημαντικές ψηφοφορίες να έχουμε και πάλι την ευκαιρία να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων και ίσως να κάνουμε και κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με, αυτό που κάνουμε εδώ. Ε, στο παρελθόν ασχοληθήκαμε πολύ αποφασιστικά με την, κατάσταση, την εξής κατάσταση στο Συμβούλιο όσον αφορά τα έγγραφα τα οποία χρειαζόμαστε την απαλλαγή δεν τα έθεσε στη διάθεσή μας και αντιδράσαμε σε αυτό και με την ομάδα εργασίας μου ε, στήριξα αυτό τον τρόπο εργασίας γιατί υποστηρίζω την νομική άποψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της απαλλαγής και βάσει του κανονισμού της συνθήκης έχει το δικαίωμα να χορηγεί αυτή την απαλλαγή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να δεχθούμε την άρνηση του Συμβουλίου. Ε, στη σημερινή ψηφοφορία θα υποστηρίξουμε τον συνάδελφο κύριο Ριβελίνη όσον αφορά την πρότασή του να μην χορηγήσει απαλλαγή στο Συμβούλιο. Αλλά στις συνεδρίες των συντονιστών ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε ε, και να αφήνουν τους συναδέλφους των άλλων πολιτικών ομάδων. Έχουμε μια πρόταση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο είπε ότι όσο δεν θέλουμε να ορίσουμε κάποια ομάδα διαπραγμάτευσης, δεν πρόκειται να αποφανθεί επί του θέματος αυτού. Έχουμε κάπως διαφορετικές απόψεις εντός της Επιτροπής όσον αφορά το πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόταση του Συμβουλίου. Δηλαδή υπάρχει η θέση να μην διαπραγματευτούμε και η θέση να συζητήσουμε τις διαδικασίες. Και στο παρελθόν εγώ ήδη είπα ότι υποστηρίζω να συζητήσουμε επί της διαδικασίας. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι, εάν έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και πάλι, ε, αν όχι στο πλαίσιο της Επιτροπής, τότε μεταξύ των συντονιστών, αλλά θα ήθελα πραγματικά να επηρεάσουμε και τις άλλες πολιτικές ομάδες, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια σκέψη για το κατά πόσο θέλουμε να δεχθούμε αυτή την πρόταση διαπραγμάτευσης. Εγώ, όπως σας είπα, θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι σωστό και πριν ε, πάμε στην Ολομέλεια σε μια οριστική απόφαση θα πρέπει να δούμε, ε, να δούμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτής της πρότασης διαπραγμάτευσης. Η κυρία Γκρέσλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Το Συμβούλιο δεν απάντησε 32 ερωτήσεις, εμείς χρειαζόμαστε απαντήσεις, άρα δεν ε, χρειάζεται να διαπραγματευτούμε κατά πόσο χρειαζόμαστε αυτές τις απαντήσεις. Σαφώς και τις χρειαζόμαστε. Δεν μου είναι ξεκάθαρο γιατί θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Γιατί ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να καταλήξουμε μια συμφωνία κυρίων. Εγώ είμαι πολέμιος αυτής της πρότασης. Ε, όσο δεν έχουν απαντηθεί οι ερωτήσεις όλα θα πάνε την κανονική τους ε, πορεία και από τη δική μας ε, οπτική γωνία δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί απαλλαγή. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα τρόπο να παρακαμφθεί η ανάγκη απάντηση των δικών μα ερωτήσεων. Θα ήθελα να το πω και πάλι ξεκάθαρα. Όλα, όλα τα υπόλοιπα θα ήταν επιζήμια. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να διοργανώσουμε σε διάφορε προποθέσει, αν το είχε. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και δεν έχουμε άλλη λύση. Και στη συνέχεια ίσως μπορούμε να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε μελλοντικά τις διαδικασίες χωρις απαλλαγη στο Συμβούλιο. Ε, Κύριος ε, Τσαρνίκη, να ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε η Ingeborg ε, Γκρέσλε. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να επιμείνουμε εδώ πέρα. Δεν ε, ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι δεν θέλαμε να μιλήσουμε με το Συμβούλιο. Τις προσκαλέσαμε επανειλημμένα. Το Συμβούλιο δεν ήθελε να μιλήσει μαζί μας. Οπότε δεν είναι ζήτημα απλά του εάν θέλουμε να συνομιλήσουμε ή όχι. Είναι το τι τίθενται όροι για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουν οι συνομιλίες και ποιο θα πρέπει να είναι το αντικείμενό τους. Θα ήθελα λοιπόν εδώ πέρα να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για την γνωμοδότησή τους γιατί ε, μας δείχνει το πώς ε, μπορεί να προχωρήσουν τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη θα πρέπει τα ερωτήματα τα οποία αρνείται να απαντήσει το Συμβούλιο πρέπει να τα θέσουμε στην Κομισιόν στη διαδικασία απαλλαγής και μετά η Κομισιόν θα πρέπει να μας ε, ενημερώσει για το αν θα απαντήσει ε, κάτι τέτοιο. Ε, θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα ή αν ε, θα μας πει πως είναι δουλειά του Συμβουλίου. Είναι λοιπόν σαφής η θέση μας και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει αυτή τη στιγμή αν θέλει να συνομιλήσει μαζί μας το Συμβούλιο. Εμείς είμαστε πάντα διατεθειμένοι. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση. Αλλά πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρως με τους δύο τελευταίους ε, συναδέλφους. Πράγματι δεν μπορούν να αποφύγουν ε, την απάντηση αυτών των ε, ερωτήσεων θα πρέπει νομίζω να επιμένουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σοντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εκ νέου να εκφράσω κάποια δυσφορία που αισθάνομαι σε σχέση με αυτό το θέμα. Γιατί έλαβα γνώση των αναλύσεων των νομικής υπηρεσίας και ειλικρινά δεν διαλευκάνουν, δεν έχουν πολύ φως στην υπόθεση. Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε τη νομική βάση επί της οποίας η Επιτροπή ελέγχου του προπολογισμού, άρα λοιπόν το Κοινοβούλιο ασκεί το έργο της. Γιατί προτείναμε να γίνει μια ψηφοφορία Δηλαδή έχουμε την αρμοδιότητα να χορηγήσουμε την απαλλαγή ή όχι. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα νομικής αξιοπιστίας από τη μία και πολιτικής αξιοπιστίας επίσης από την άλλη. Άρα όμως ο ρόλος κάθε κοινοβουλίου σε κάθε δημοκρατία είναι να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία και να κάνει τον έλεγχο της ε, δημοσιονομικής εκτέλεσης των δημοσίων κονδυλίων και διαρωτώμε κατά πόσο εμείς ε, ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία. Γιατί. Ε, τι γίνεται εδώ, υπάρχει ένα συμβούλιο το οποίο είναι απρόθυμο, το οποίο δεν έχει ένα φυσιολογικό διάλογο μαζί μας και αυτό προκαλεί εκνευρισμό στους ε, βουλευτές που έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Αλλά τι παρατηρούμε, παρατηρούμε ότι στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, που είναι ο βραχίωνας ε, του Κοινοβουλίου. Έχουμε 350 σελίδες ε, παρατηρήσεων ε, κατά της Επιτροπής και παρόλα αυτά χορηγείται απαλλαγή. Ενώ δεν αναφέρεται τίποτα για το Συμβούλιο και εμείς θέλουμε να μην τους δώσουμε την απαλλαγή. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο να μας εξηγήσει και ενδεχομένω να στήσει μια αποστολή στο Συμβούλιο. Και αν δεν το πράξει αυτό το ελεγκτικό συνέδριο, τότε στην περίπτωση αυτή γιατί δεν θέλουμε να συστήσουμε μια εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου για τις δραστηριότητες του Συμβουλίου, ώστε να έχουμε μια νομική βάση για να δούμε και μια ισχύ, εξουσία μάλλον, για να δούμε τι γίνεται στο Συμβούλιο γιατί ε, αν διαβάσουμε τη συνθήκη, όλα αυτά συνδέονται με τον κανονισμό και νομίζω δεν υπάρχει νομική βάση για να χορηγήσουμε εμείς ε, την απαλλαγή σε κάποιο θεσμικό όργανο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία χορηγεί την απαλλαγή, Ενδεχομένω η Κομισιόν, αλλά ίσως να απατώμε. Δεν ξέρω. Ήδη έχω εκφράσει αυτή μου την άποψη. Ο κύριος Κυλακάκης έχει το λόγο. I uh, uh, Και εγώ θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι το Συμβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το Συμβούλιο αποφεύγει να σχολιάσει τις θέσεις μας και μας αγνοεί εδώ και καιρό. Πρέπει λοιπόν με ηρεμία αλλά και επιμονή να συνεχίσουμε την πορεία μας. Κυρία Γκρέσλε. Συγγνώμη που παίρνω πάλι τον λόγο. Δεν θα ήθελα βεβαίως εδώ πέρα να διαφωνήσω με τον Ζαν Πιεροντή, αλλά κοιτάξτε, αναρωτιέμαι ώρες ώρες, ε, καταλαβαίνω πως είναι διαφορετικές οι παραδόσεις για το κατά πόσον είναι δημοκρατία η Γαλλία, γιατί βεβαίως οτιδήποτε είναι ε, προϋπολογισμός προπολογισμό Ένωση αφορά την Επιτροπή μας. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στον ε, κανονισμό. Και απλά θέλω να Ε, τηρηθούν αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε την εντύπωση πως αμφιβάλλουμε για το ορθό και την νομιμότητα ε, των όσων κάνουμε. Οπότε εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι είναι πράγματι υποχρεωμένο να μας δέσει αυτές τις πληροφορίες στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος τον λόγο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ριβελίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από οτιδήποτε άλλο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους γιατί πέρα από την πολιτική τους τοποθέτηση οι περισσότεροι από εμά βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, παρουσιάζεται σαν εκπρόσωπος των πολιτών που το εκλέγουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πέραν των πολιτικών πεπιθήσεων και τοποθετήσεων του καθενός εμένουμε στον σεβασμό συγκεκριμένων αρχών όλοι μαζί. Η δεύτερη παρατήρηση είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Δεν πήραμε τις σωστές απαντήσεις από το Συμβούλιο, είναι σαφές. Και η νομική υπηρεσία στην ουσία εξέδωσε μία γνωμοδότηση σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα της νομοδότησης της νομικής υπηρεσίας λέγει ότι με το κλείσιμο των λογαριασμών και την απαλλαγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε όπως λέει το 219 της συνθήκης το τεχνικό κομμάτι της απαλλαγής. Η νομική υπηρεσία όμως μας υποστηρίζει και ανοίγει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όταν αναφέρεται στην πολιτική σημασία της δικής μας γνωμοδότησης και αυτό κάνουμε εμείς στην ουσία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε οδήποτε δισταγμό σήμερα, θα πρέπει να εμείνουμε στην πορεία μας. Γιατί αν θέλετε και σε τεχνικό επίπεδο από πλευράς της νομικής υπηρεσίας υποστηριζόμεθα και θεωρείται σωστή η αντιμετώπιση μας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Καταρχάς πρόταση απόφαση στο σύνολό της είναι υπέρ παρακαλώ. είναι κατά αποχή κανείς, γιατί ομόφωνα... Α, υπάρχει μία αποχή. Συγγνώμη, μαθαίνω, δεν τα έχω μάθει καλά. Μία αποχή λοιπόν. Συνεπώς γίνεται δεκτή ομόφωνα με μία αποχή μάλλον. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω στην παράγραφο 5 την προφορική τροπολογία α. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές μία αποχή πάλι δεκτή. Παράγραφος 6 προφορική β ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 7 προφορική γ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές Δεκτή με μία αποχή. Παράγραφος 8. Προφορική δέλτα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο κατά μία αποχή δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία 3 μάλλον η οποία έχει καταπέσει, η 9 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές μία αποχή δεκτή η πέντε έχει αποσυρθεί έχω την τροπολογία ένα εδώ ποιοι είναι υπέρ της ένα ποιοι είναι κατά τέσσερις κατά δεκτή Στην αιτιολογική σκέψη Γ έχω την τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Δεν γίνεται δεκτή η τροπολογία 2 και τώρα ψηφίζουμε το τροπολογημένο ψήφισμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι πλέον ομόφωνα γίνεται δεκτή. Τα συγχαρητήριά μου κύριε Ριβελίνη. Α, έπρεπε να μετρήσω τη ψηφοφορία. Γι' αυτό λοιπόν μια φορά ακόμα. Ποιοι είναι υπέρ. Ξαναψηφίζουμε. Πρέπει να μετρήσω τις ψήφους. Δεν το ξέρω. Ευχαριστώ. Επιβεβαιούται λοιπόν δεκτή. Τώρα, Περνάμε στο 4 της ημερήσιας διάταξης για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Ο εισηγητής θέλει να μας πει κάτι ή κάποιος άλλος. Δεν έχω κάτι να προσθέσω, λέει ο κ. Σταυρακάκης. Θέλει κάποιος να κάνει άλλη παρατήρηση. κύριε Ανδρέασεν, να πω ότι ίσως είμαι η μόνη βουλευτής εδώ η οποία έχει επισκεφθεί το αστυνομικό κολέγιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είδα ότι πράγματι κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να βελτιώσουν τα πράγματα και δίνουμε απαλλαγή στον προϋπολογισμό του 2009 της Ακαδημίας αυτής είχαν διαχειριστεί τα πράγματα τότε αυτοί για τους οποίους ε, είχαν, από τους οποίους είχαν διαπρακτεί μη κανονικές ενέργειες και γι' αυτό θα καταψηφίσω α, τις, πρότασεις, αυτές. Και αν εγκρίνουμε τις προτάσεις αυτές ε, νομίζω ότι δεν θα προσφέρουμε τίποτα στη νέα διαχείριση της Ακαδημίας αυτής. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο? Όχι κυρία Γκρέσλε, συγγνώμη. Ε, δεν είναι αλήθεια ότι εδώ είναι οι καλοί που δεν θέλουν να χορηγήσουν επαλλαγή και οι κακοί από την άλλη. Ε, ε, θα ήθελα να συγχωρέσω την κυρία Μάρκοβα γιατί βρίσκεται στι Ηνωμένε Πολιτείε, διδάσκει εκεί αυτή τη στιγμή και λέει ότι θα παίρναμε ε, πολλά έγγραφα από τον Οργανισμό Φαρμάκων κυρίως. Αλλά τελικά δεν τα πήραμε αυτά που θέλαμε. Ε, ε, νομίζω ότι πράγματι και οι δύο αυτοί οι οργανισμοί έχουν βελτιώσει τη διαχείριση, έχουν διανύσει μια μακρά πορεία. Γι' αυτό ίσως το 2010 πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε όλη την ιστορία με το θάρρος που έχει επιδείξει η κυρία Μάρκοβα. Να το τονίσουμε αυτό, γιατί πραγματικά έχω εμπιστοσύνη ότι το 2010, εν πάση περιπτώσει, θα μπορέσουμε να διαπιστωθούμε να διαπιστώσουμε τότε κατά πόσα έχουν γίνει πράγματι, έχουν εμπεδοθεί αυτές οι βελτιώσεις. Νομίζω θα πρέπει δηλαδή, να στραφούμε στο 2010. Μάλιστα. Δεν θέλει, φαντάζομαι κανείς άλλος να μιλήσει, οπότε περνάμε στην ψηφοφορία. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα για το εκτιμώντα 11α τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μια αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Μετά ψηφίζουμε την πρόταση επί της απόφασης στο σύνολό της. Ποιος είναι υπέρ. Ε, αν έχετε τις κάρτες ε, μαζί σας. Για να μην κάνουμε γυμναστική, μπορούμε να ψηφίσουμε με τις κάρτες. Άρχεται τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Όχι. Ωραία, το λαμβάνουμε υπόψη. Πέρας της ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα είναι 16 υπέρ και 14 υπέρ. 2 κατά. Συν. Ο κύριο Γκάιερ 15 υπέρ. Άρα γίνεται δεκτή. Πρέπει να τα μάθουμε. Καταλαβαίνετε. Οπότε γίνεται δεκτή. Μετά έχουμε την πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών. Ποιο είναι υπέρ. Επίση επίσης με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. ψήφισαν όλοι. Πέρας. Η μηχανή δουλεύει. Δηλαδή. Ε, η ψήφος μου δεν καταγράφηκε γιατί δεν ε, μπόρεσα να φτάσω στο μηχάνημα κύριε Πρόεδρε. Σα μετρήσαμε ούτω ή άλλω υπέρ, οπότε 15 υπέρ είχα πει ούτω ή άλλω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε λοιπόν. Στο σχέδιο ψηφίσματος παράγραφος 1, τροπολογία 2 υπέρ. Νομίζω πως η πλειοψηφία είναι υπέρ. Παράγραφος 1 CA. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 1α νέο. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 1β, νέα, τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως η είναι υπέρ. Τροπολογία 1 γάμα νέο. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. πέντε βλέπω. Κατά, άρα γίνεται δεκτή. Παράγραφος 1 δέλτα νέο, τροπολογία 7. Α, έχει αποσυρθεί μάλιστα. Παράγραφος 2, τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. 3 κατά, μία αποχή δεκτή. Τροπολογία 3. Τροπολογία 9, με συγχωρείτε, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω πως η πλειοψηφία είναι υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ωραία, να επαληθεύσουμε. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν 8 υπέρ 6 κατά 2 αποχές. Τροπολογία 4, ναι, παράγραφος 4, τροπολογία 10, με συγχωρείτε, Ποιο είναι υπέρ. Θέλετε το λόγο, κύριε Γκάιρ. Εμένα πρέπει να με μετρήσετε στις ψήφους ε, κατά, οπότε το αποτέλεσμα είναι 8 έναντι 7. Μάλιστα, με συγχωρείτε. Δεν ε, τα καταφέραμε. Λοιπόν, Τροπολογία 10, ποιος είναι υπέρ. Νομίζω πως είναι η πλειοψηφία, υπάρχει τουλάχιστον ένας κατά. Παράγραφος 7, τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Μάλλον γίνεται δεκτή. Παράγραφος 7α. Νέο. Τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω τρεις. Κατά. Άρα γίνεται δεκτή. Παράγραφος 9. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Κανείς. Άρα ούτε αποχές. Οπότε υποθέτω πως γίνεται δεκτή. Παραγραφός 14, τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Γίνεται λοιπόν δεκτή. Παράγραφος 15, τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κανείς δεκτή. Παράγραφος 18, τροπολογία 16 υπέρ. μετά αποχές δεκτή. Οπότε ψηφίζουμε για το σχέδιο ψηφίσματος στο σύνολό του ηλεκτρονικά και την ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Το αποτέλεσμα είναι σαφές 15 υπέρ και μία κατά, άρα γίνεται δεκτό. 16 του κυρίου Γκάιρ συμπεριλαμβανομένου. Οπότε τελειώσαμε το σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη και περνάμε στο 5ο. Απαλλαγή της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων. Καμία παρατήρηση από τον συγκητή. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Όχι. Περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Πρώτος η απόφαση για την απαλλαγή λοιπόν. Έχουμε την τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Αποχή. Και μία αποχή. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχή ένας κατά μία αποχή δεκτή τροπολογία 1 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές μία αποχή δεκτή ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για την πρόταση απόφαση στο σύνολό της άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 2 αποχές. Δεκτή. Και ο κύριος Γκάγερ ένας 15 υπέρ. Τώρα για το κλείσιμο των λογαριασμών. Παράγραφος 1, τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Δεκτή. Παράγραφος το απολογια 5 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Δεκτή. Τώρα ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραστη ψηφοφορία. 14 υπέρ, 2 αποχές. Η πρόταση απόφασης γίνεται δεκτή. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα. Τροπολογία 6. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. κατά αποχές ένας κατά μία αποχή δεύτερο τμήμα είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Επτά υπέρ, νέα κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Και εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε την 7. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. 9 υπέρ 6 κατά. Συνεπώς γίνεται δεκτή. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Τις 8. Κατά. Και εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 8. Ψηφίζουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες Ο κύριος Γκάγερ αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά. 9 υπέρ, 8 κατά. 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Δεν υπάρχουν αποχές δεκτή. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ της 10. Ποιοι είναι κατά της 10. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 11 καταπίπτει. Τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές με τρεις ψήφους κατά γίνεται δεκτή. Τροπολογία 13. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή 13. 14 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά αποχές τρεις κατά δεκτή 15 κατά πίπτη 16 ποιοι είναι υπέρ Α, συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε τη δεκαπέντε, λάθος. Ψηφίζουμε την δεκαπέντε λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά της δεκαπέντε, Απέχουν Δεκτή. Η 16 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές με τρεις κατά γίνεται δεκτή. 17 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 18. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 19 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 20 τροπολογία. 20 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές με τρεις ψήφους κατά γίνεται δεκτή. Τροπολογία 21. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 21 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα έχουν όλοι κάρτες. Πέρα της ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι 10 υπέρ 7 κατά. Συνεπώς δεκτή. Παράγραφος 14 τροπολογία 22 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22 ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή 9 υπέρ 8 κατά. Λοιπόν, 23. Ποιοι είναι υπέρ της 23. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Με τρεις ψήφους κατά. 24. Ποιοι είναι υπέρ της 24. Κατά. Αποχές. Δεκτή 24. Και στο τέλος το σύνολο του ψηφίσματος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 16 υπέρ. Μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε εισηγητά. Το επόμενο θέμα, ο εξυγχρονισμός των τελωνίων. Ο εισηγητής θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, τέσσερις ε, τροπολογίες έχουν κατατεθεί για αυτή τη γνωμοδότηση. Στις τρεις από τις τέσσερις ε, μπορώ να συμφωνήσω. Με την πρώτη μόνο του Ρολάντα Πάξας ε, ε, διαφωνώ γιατί δεν καταλαβαίνω την ε, τροπολογία, είναι μεταφρασμένη στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες και δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ο κύριος ε, Πάξας. Προσπαθήσαμε να το δούμε στο πρωτότυπο, αλλά ούτε και εκεί πέρα μπορούσε να με βοηθήσει η γραμματεία. Οπότε μπορεί βεβαίως να διορθωθεί αργότερα αυτή η κατάσταση, αλλά προς στιγμή είμαι κατά αυτής της τροπολογίας. Θα ήθελα να πω μόνο πως ε, ε, έχουμε, θα έχουμε μια μετάφραση σήμερα. Έχουμε λοιπόν τις, δύο ε, τις δύο και τρία στις οποίες υπήρχε ένα πλήν. Από όταν έδωσα λοιπόν την μετάφραση είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα και άρα το ΕΛΚ συμφωνεί με τον συγητή. Κύριε Πρόεδρε, μας δυσκολεύουν τα πράγματα εδώ πέρα με τις ε, μεταφράσεις. Ε, είμαστε δημοκρατικά οργανωμένοι, πρέπει να μπορούμε να συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Ε, η τελευταία μας συνεδρίαση ήταν την τρίτη που μας πέρασε στο Στρασβούργο. Έχουμε εδώ και καιρό λοιπόν τη γνωμοδότηση, αλλά οι τροπολογίες δεν είχαν μεταφραστεί. Θα ήθελα να παρακαλέσω να ξαναδούμε αυτό το σημαντικό θέμα για να μπορούμε να συζητήσουμε μεταξύ μας. Δύο φορές το έχουμε βάλει στη μερίσια διάταξη και δεν έχουμε μπορέσει να το συζητήσουμε. Πρέπει να το ξαναδεί η γραμματεία. Ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία, αν δεν έχει κάποιος άλλος καμία παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα παράγραφος 2 τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Με μία αποχή, από όσο βλέπω, απορρίπτεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω καλό είναι να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 2, παράγραφος 3. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Γίνεται λοιπόν δεκτή. Παράγραφος 3α, τροπολογία 3, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 5α, τροπολογία 4, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Με μια αποχή. Δεκτή. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης, ηλεκτρονικά αρχή ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 16 υπέρ. Μια ψήφο κατά. Τα συγχαρητήριά μου στον Αντιπρόεδρο. we... Το, τώρα θα περάσουμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης που είναι ο δημοσιονομικός έλεγχος της χρηματοοικονομικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Κύριε Γκάιερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως ε, ε, σήμερα είμαι μόνος εμψυχωτής σε αυτή την ε, επιτροπή αλλά θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, όσον αφορά αυτή την έκθεση πρωτοβουλία για, για την συνδρομή στο Αφγανιστάν, για τον έλεγχο της υποστήριξης του Αφγανιστάν, θα ήθελα να σας πω ότι ο συνάδελφος Πίνο Λάκη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη δική του έκθεση πρωτοβουλίας υπέβαλε μια νέα πρόταση για μια ευρωπαϊκή στρατηγική στο Αφγανιστάν. Και σε σχέση με την έκθεση αυτή, ε, προσέκρισε σε κάποιες ε, παρατηρίες που αφορούν, τα σταλίες που αφορούν τη χρήση των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων στο Αφγανιστάν. Και εξού λοιπόν και ζητήθηκε μία έκθεση πρωτοβουλίας και εγώ είχα τη χαρά να γράψω ένα σχέδιο έκθεσης. Και πρόκειται για μία μαδική εργασία ε, η οποία έγινε, συστάθηκε η ομάδα αυτή με τη βοήθεια της ε, γραμματείας, την οποία ήθελα να ευχαριστήσω, καθώς και στον βοηθό μου. Και πολύ γρήγορα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έχει νόημα να εξετάσουμε ε, ποιο δρόμο ακολουθούν τα χρήματα για να φτάσουν στο Αφγανιστάν και ποια είναι τα ειδικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διάβολων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κονδύλια αυτά. Εάν ασχοληθούμε με αυτούς που είναι αρμόδιοι για τη δίκηση αυτών των διάβλων, ε, καταλήγουμε σε ορισμένα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνεπάγονται τα κανάλια αυτά, αυτή η διάβλη. Δηλαδή, και ε, όσον αφορά τις πληροφορίες για αυτούς τους διάβλους, ε, πήραμε πολύ βοήθεια ε, στην εξέταση των ε, προγραμμάτων τα οποία υλοποιούνται στο Αφγανιστάν εκ μέρους των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση εδώ που ίσως δεν σημαίνει όλοι οι συνάδελφοι στην Επιτροπή. από την άλλη πλευρά Ίσως δεν μπορούμε να σημειώσουμε πραγματικά βήματα πρόοδου στη χώρα αυτή στο Αφγανιστάν εάν η διοίκηση στο Αφγανιστάν όσο και στοιχειώδης να είναι οι διαδικασίες της δεν βοηθηθεί να φτάσει σε ένα σημείο τελικά η ίδια που ε, να έχει μια υπεύθυνη διαχείριση των χρημάτων των διεθνών ε, δωρητών. Να εκμάθει αυτή τη διαδικασία και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διατρέξουμε ορισμένου κινδύνου, να πάρουμε κάποια ρίσκα. Οι Αμερικανοί που το δοκίμασαν ε, πλήρωσαν πικρά γι' αυτό. Ήταν μια πικρή εμπειρία αυτή για τους Αμερικανού. Και όταν κάναμε μια έρευνα στο πλαίσιο της έκθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί ακούσαμε διάφορες ιστορίες ε, για το τι έμαθαν οι διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες όσον αφορά τη χρήση αυτών των κονδυλίων. Και υπάρχει μια γλαφυρή τεκμηρίωση της χρήσης αυτών των χρημάτων. Ε, για παράδειγμα, τα ρευστά έφτασαν σε χαρτόνια στο Αφγανιστάν, σε κυβότια, ε, και μόνο ένα μέρος αυτών των χρημάτων. Η καλή είδηση είναι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια όσο εγώ μπορούσα να διαπιστώσω δεν ήταν μεταξύ αυτών των χρημάτων. Δηλαδή, εμείς ε, τα χρήματα δικά μας πήραν ε, ένα ασφαλή δρόμο και δεν έφυγαν από τη χώρα όπως τα αμερικάνικα χρήματα που τελικά φύγαν μέσα σε αυτά τα χαρτοκιβώτια. Τώρα, όσον αφορά το λεγόμενο capacity building, ε, τη δυνατότητα δηλαδή να υποστηριχθούν οι αφγανικές αρχές για τον αποτελεσματικό χειρισμό αυτών των κονδυλίων, για την αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων ε, και για το πώς μπορεί κανείς να καταμετρήσει αυτά τα αποτελέσματα. Είναι ένα στόχος ο οποίος πραγματικά θα πρέπει να υποστηριχθεί εκ μέρους μας γιατί είναι ένα βιώσιμο στόχος. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή την κατάσταση, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν τη στιγμή που ε, θα αποσυρθεί όχι μόνο ο στρατός αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, και ήδη το έχουν πράξει σε μεγάλο βαθμό. Για να υποβοηθήσουμε λοιπόν την οικοδόμηση των υπηρεσιών σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση των υπηρεσιών. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, οι ανησυχίε μας θα αυξηθούν για το τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, θα πρέπει ε, να δούμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους του Αφγανούς να οικοδομήσουν αυτές τις δομές. Το capacity building δηλαδή οι γνωμοδοτήσεις οι οποίες ε, συντάχθηκαν από την ΑΦΕΤ και την ΤΕΒΕ πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και όλα αυτά κινούνται και στην ίδια γραμμή που έχει κινηθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει λάβει αποφάσεις μέσω των εκθέσεων αυτών των δύο επιτροπών. Ε, είναι λοιπόν μια διαδικασία που έχει βρει υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είναι και μια διαδικασία για την οποία θα πρέπει να συμφωνήσουμε και εμεί ήδη, γιατί ενδεχομένω εμείς τη θεωρούμε αμφίβολη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει επακριβής έλεγχος και θα πρέπει να διατυπώσουμε επακριβείς και αυστηρές ε, προδιαγραφές για την άσκηση του ελέγχου. Ε, για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε τη χορήγηση άμεσης ε, βοήθειας στο Αφγανιστάν οι Αμερικανοί υπήρξαν αρχικά πολύ αφελείς όπως σας το είπα και πλήρωσαν πολύ ακριβά γι' αυτό και τώρα ακολουθούν και το δρόμο αυτό που σα προτείνω εγώ να συνδέσουν την παρχή βοήθεια με πολύ αυστηρούς όρου, και συνέγραψαν αυτή την έκθεση και όσον αφορά το Υπουργείο Υγεία, πρώτη φορά βρίσκουν την εφαρμογή του αυτοί οι κανόνε πράγματι. Ωστόσο οι κανόνε, όπω σα είπα θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και διαφανεί, Αυτό εξυπηρετεί τα δικά μα συμφέροντα, συμφέροντα τη Κομισιόν αλλά και τη Αφγανική Διοίκηση και κυβέρνηση θα πρέπει να γνωρίζουν ποιου κανόνε καλούνται να τηρήσουν. Αυτή τη στιγμή ε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση των ελεγκτικών μηχανισμών στο Αφγανιστάν. Το Αφγανικό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές με τις οποίες είμαστε εμείς εξοικειωμένοι και αυτό σχετίζεται με το ότι τα μέλη του συνεδρίου διορίζονται από τον πρόεδρο και όχι από το κοινοβούλιο. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν στο Αφγανιστάν παραμένει στα χέρια της κυβέρνησης και όχι της ε, εκπροσώπησης του λαού. Και όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν μέσω μιας ε, νομοθεσίας που αυτή τη στιγμή γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευση στη χώρα και μία από τι προποθέσει που θα πρέπει εμεί να στέλνουμε είναι το ελεγκτικό συνέδριο στο Αφγανιστάν να μην είναι εξαρτημένο από την κυβέρνηση αλλά να πληρεί διεθνείς προδιαγραφές, γιατί αυτά είναι κεντρικά σημεία που αφορούν το δημοκρατικό έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο, με το οποίο θα πρέπει να συνδεθεί η άμεση χορήγηση βοήθειας. Προσπάθησα να εξετάσω ποια είναι τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κονδύλια μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων ή μέσω trust funds ή για κονδύλια που δίνονται ως άμεσης βοήθεια στον προπολογισμό και τέλος προσπάθησα να δω τι γίνεται με τους ε, ιδιώτες εταίρους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό σημείο που θα πρέπει πραγματικά να αποφασίσουμε κάποιους ε, συγκεκριμένους κανόνες. Το σύστημα της υπεργολαβίας, του subcontracting. Ε, και υπάρχουν, ε, διαπιστώσαμε κάποιες καταστάσεις όπου για ορισμένε ιδιωτικέ συμβάσεις ε, έχουν επιλεγεί περισσότεροι εταίροι και όπου τα χρήματα ε, τα οποία θα συνέβαλαν στην οικοδόμηση του Αφγανιστάν τελικά δεν εξυπηρέτησαν αυτό το σκοπό αλλά ε, βρέθηκαν τα χέρια αυτά σε διάφορες εταιρείες ε, ανάθεση έργων υπεργολαβικές που τελικά δεν είχαν καμία σχέση με την ποιότητα των υποεξέλιξη έργων και τελικά ζημίωσαν τον πολιτικό στόχο της ενίσχυσης της αφγανικής οικονομίας. Αν υπάρχει λοιπόν ένας υπεργολάβος θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για το από πού θα πρέπει να προέρχεται και αν προέρχεται από το Αφγανιστάν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ε, να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να προτιμάται ένας Αφγανός εταίρος ε, αλλά τελικά να διανέμονται τα χρήματα μεταξύ περισσότερων μέσω μιας απάτης τελικά. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι αθέμητη και η οποία δεν εξυπηρετεί τη σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων ούτε την εξυπηρέτηση των πολιτικών σκοπών. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές προτάσεις που υποβάλλω στην έκθεση αυτή και αναμένω τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις και σχόλια. κυρία Γκρέσλε, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η σκιώδη συγγήτρια η Μόνικα Χόλμα είναι ακόμα στο αεροδρόμιο στη Γερμανία και ζητά συγγνώμη Γι' αυτό θα ήθελα να μεταφέρω τον έπαινο της. Η έκθεση είναι πολύ καλά, πολύ ισορροπημένη, με έρευνα των γεγονότων, έχει αναφέρει τα διάφορα προβλήματα. Απορίσαμε βεβαίω για το πόσο... και εκλογήκαμε από το πόσο κουράστηκε ο Γέννης, μίλησε με τους Αμερικάνους Βεβαίως ε, είναι σαφές πως ε, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό με τα συνήθη κριτήρια των Βρυξελών και άλλων ε, σημείων του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει παραδεχτεί και το ελληνικό συνέδριο σχετική του έκθεση για τα κονδύλια πάνε στον ΟΗΕ στο κεφάλαιο του Αφγανιστάν. Ένα... Κάποια ερωτήματα τώρα ποιο ρόλο παίζει η τοπική αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Αφγανιστάν, τι εμπειρίες είχες μαζί τους όσον αφορά την ε, οικοδόμηση, αν θέλετε, εκεί πέρα της διοίκησης. Ακούω φοβερά πράγματα για τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατασκευές και η λογοδοσία επίσης, το τι γνωρίζουμε τελικά δεν αλλάζει ε, το γεγονός πως ε, θα έπρεπε να υπάρξει κάποια λογοδοσία. Εμένα 29 Σεπτεμβρίου είπε στα χέρια μου ένα σημείωμα το οποίο δεν έλεγε καθόλου ευχάριστα πράγματα όσον αφορά την πρεσβεία εκεί πέρα. Οπότε το ερώτημα που θέθηκε και η είναι το εάν ο προϋπολογισμός λύνει τα προβλήματα τα οποία έχουμε γιατί βέβαια εντάξει δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να επαληθεύσουμε, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τις προσωπικές σου εντυπώσεις. Και μια συμβουλή, τι, κάνουμε με τα, τι να κάνουμε με τα χρήματα αυτά και με τα χρήματα του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν. Εγώ είμαι η συγγήτρια για την ειδική αυτή έκθεση. Γι' αυτό θα ήθελα την άποψή σου. Και όπως είπα, ε, σε εκτιμούμε για το ότι Ασχολήθηκε με αυτό το σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντάκτη της ε, γνωμοδότησης αυτής της εξαιρετικής αυτής γνωμοδότησης γιατί και ξέρετε η αμερικανική εμπειρία ε, αναφέρθηκε και όπως αναφέρει και ο εισηγητής εδώ πέρα, η αμερικανική προσέγγιση στην αρχή ήταν κάπως αφελής. Τι σημαίνει αυτό. Για τις εκατομμύρια δολάρια έφταναν στο Αφγανιστάν και κατέληξαν σε τράπεζες στην Ελβετία και στη Σαουδική Αραβία. Και ποιος ξέρει πού. Οπότε το ερώτημα το οποίο θα ήθελα και εγώ να κάνω μετά από αυτά τα οποία είπε και η Ίγκεμπορκ Κρέσλε είναι εάν είναι δυνατόν να ακούσουμε λίγα πράγματα περισσότερο, περισσότερα. Δηλαδή, είναι σε θέση η αυγανική διοίκηση να αποδεχτεί βοήθεια στον προπολογισμό, γιατί είναι ένα πράγμα είναι να θέτουμε εμεί απαιτήσει και κριτήρια μετρήσιμα, αλλά το θέμα είναι εάν δούμε την αυγανική διοίκηση ως έχει αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα προϋπολογισμό και μια βοήθεια. Any other Κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε το λόγο. Η Επιτροπή θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Δεν έρχομαι συχνά εδώ. Είμαι υπεύθυνο για την Ασία και για τη συγκεκριμένη χώρα για το Αφγανιστάν. Θα είμαι σύντομος. Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις συστάσεις τις οποίες κάνει. Δεχόμαστε τις περισσότερες από τις συστάσεις αυτές απόλυτα. Κάποιες από αυτές βέβαια θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο για να τις κατανοήσουμε κάπως καλύτερα. Θα ήθελα επίσης να κάνω λίγες παρατηρήσεις σχετικά με την μεταφορά των στοιχείων του προϋπολογισμού. Έχει τεθεί το θέμα αυτό επανειλημμένα στο παρελθόν. Εμείς δεν υποστηρίζουμε καταρχάς τα δημοσιονομικά του Αφγανιστάν άμεσα. Εμείς δίνουμε τα λεφτά στον προϋπολογισμό και οι αφγανικές αρχές να είναι υπεύθυνε για τη διάθεση των χρημάτων αυτών. Δεν το κάνουμε αυτό. Απαιτούμε όμως διάφορους δημοσιονομικούς στόχους όπως τη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως επίσης και τα συστήματα μικροδιαχείρισης, τα δημοσιονομικά, αλλά αυτά δεν είναι σε ενέργεια στο Αφγανιστάν. Εμπλεκόμεθα σε τομείς όπως η υγεία, η γεωργία, η ανάπτυξη της υπαίθρου. Υπάρχει μια βελτίωση, υπάρχει καλή συνεργασία με τα εθνικά επίπεδα και το τέταρτο τομέα είναι η ασφάλεια. Όσον το θέμα της ασφάλειας δεν βελτιώνεται στο Αφγανιστάν και μάλιστα τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες χειροτερεύει η κατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά την οποία θέλουμε. Ξέρετε ότι για μικρό χρονικό διάστημα οι συνάδελφοι ε, που εργάζονται εκεί δεν μπορούν να βγουν από το κτίριό τους ε, αν δεν τους δοθεί ειδική άδεια εμείς ας πούμε από την ΤΕΦΚΟ, τη Γενική Διεύθυνση, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε επί τόπου και να παρακολουθούμε την εφαρμογή των προγραμμάτων. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, συνεπώς θα απαιτηθεί πολύ χρόνος έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε τους στόχους μας αυτούς ε, μέσω άμεσης δημοσιονομικής στήριξης. Προσπάθειες γίνονται όπως ξέρετε σε συνεργασία και με άλλους δωρητές, ε, με την Παγκόσμια Τράπεζα, όπως επίσης και το πρόβλημα τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών και την αστυνομική δύναμη Εμείς υποστηρίζουμε τη δημιουργία των ανοιχτών δημοσιονομικών συστημάτων τις οποίες θέτουν σε λειτουργία οι αφγανικές αρχές έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν σωστά τους δικούς τους δημοσιονομικούς κανόνες και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό μέσω των συγκεκριμένων διαπιστευμάτων που λειτουργούν σαν ασφάλεια. Και δεν υπάρχει πληρωμή αν δεν αδειοδοτηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια είτε από την διαχειρίστρια υπηρεσία είτε από την Παγκόσμια Τράπεζα. Θα θέλαμε όπως σε άλλες χώρες να περάσουμε σε απευθεία στήριξη μέσω του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε σχετικά γρήγορα, όπως και με άλλες χώρες της Ασίας, αλλά στο σημερινό πλαίσιο, στο Αφγανιστάν, με τη συγκυρία η οποία επικρατεί, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Τώρα, για τη νέα αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ο διορισμός του κυρίου Βιγκόντας, ειδικού εκπροσώπου και ο νέος ρόλος της ε, Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας από την 1η Ιανουαρίου του 2011 έχει βελτιώσει κατά πολύ τον ρόλο μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περισσότερο ορατή επιτόπου από ό,τι στο παρελθόν. Ο πρέσβης λειτουργεί με συντονιστικό τρόπο ανάμεσα στις διάφορες χώρες της Ένωσης και όλο και περισσότερο δίνουμε ένα καλό παράδειγμα προς τις υπόλοιπες χώρες, όχι τέλειο. Υπάρχουν όμως ε, σαφέστατα ε, χώρια βελτίωση. Και αυτό φαίνεται και στα ετήσια προγράμματα δράσης, τα οποία συνυπογράφουμε σαν Επιτροπή και κράτη-μέλη. Θα πρέπει τα προγράμματα αυτά δράσης να μπορέσουν να σφραγίσουν την αγαστή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και μέσω των εφαρμοστικών εκθέσεων σε επίπεδο τοπικό. Κυρία Γκρέσλα. Ναι, όταν λέτε ότι υπάρχουν βελτιώσεις, πού υπάρχουν οι βελτιώσεις και τι έπρεπε να βελτιωθεί. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Τι έχριζε βελτίωσης. Έπειτα ο πρέσβης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ζήτησε να τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας μιας, ε, ενός χώρου γκολφ. Τι άλλο έκανε. Επίσης τι συμβαίνει με, το, με τη δημιουργία ενός σχολείου το οποίο είχε προταθεί. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ο Γιάννης Γκάιερ θα απαντήσει στο ερώτημά μου και το ομολογώ ανοιχτά ενέχεται η πρόθεση να δώσουμε στους συναδέλφους της Κομισιόν την ευκαιρία να μας πούν πώς μπορούν να ελεγχθούν τα προγράμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Αφγανιστάν. Κάναμε μια σχετική συζήτηση και στην πρώτη μου παρουσίαση, ωστόσο δεν ε, θέλησα να αναφερθώ στο έργο της Κομισιόν Επιτόπου στο Αφγανιστάν. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να πούμε άλλη μια φορά εδώ στην Επιτροπή με ποιο τρόπο η Κομισιόν ελέγχει την ε, εκτέλεση προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται στο Αφγανιστάν. Θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει κανείς άλλος ο οποίος θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Η Κομισιόν να απαντήσει. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο τρόποι εφαρμογή υπάρχουν στην Αφγανιστάν. στο Αφγανιστάν. Πρώτα απ' όλα η κοινή διαχείριση. Γύρω στο 300-400 εκατομμύρια από τα προγράμματά μας πάνε μέσω δύο καταπιστευμάτων τα οποία έχουμε και χρησιμοποιούμε το, τα συστήματα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και όπως σας εξήγησα πριν από λίγο, ε, φαίνεται εκεί πέρα κάθε έξοδο που υποβάλλουν για πληρωμή οι αρχές. Οπότε η εγγύηση όσον αφορά τον κίνδυνο προέρχεται από την Παγκόσμια Τράπεζα αφενός και αφετέρου από την Λότφα. Και η δεύτερη πτυχή είναι μια κεντρική διοίκηση, δηλαδή η δική μας η αντιπροσωπεία κάνει και τις αναθέσεις και τις ε, πληρωμές σε ΜΚΟ στις οποίες αναθέτει. Κατά κανόνα προσπαθούμε να συνεργαστούμε με γνωστές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ομολογώ βεβαίω πω εκεί πέρα ο κίνδυνο είναι κάπω υψηλότερο και βέβαια το πρόβλημα που έχουμε ειδικά για την κεντρική αυτή διαχείριση είναι πω δεν μπορούμε να επιβλέψουμε επιτόπου. Δεν μπορούμε να πάμε επιτόπου να δούμε τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται. Κατά κανόνα χρησιμοποιούμε ντόπιου. Αλλά ακόμα και σήμερα οι ντόπιοι δεν επιτρέπεται να πάνε επιτόπου στι επαρχίε για να παρακολουθήσουν τα έργα αυτά γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Ελπίζουμε αυτή η κατάσταση να μην διαρκέσει. Σας ευχαριστώ. Παρατηρήσεις. Η κυρία Γκρέσλε. Ναι, το περίμενα. Δηλαδή, για να το πω εγώ απλά, δεν ξέρουμε ε, τίποτα. Δεν προξενεί έκπληξη και πριν από δύο χρόνια είχαμε κάνει μια έκθεση δύο πρωτοβουλία για το Αφγανιστάν. Ήταν και ο συνάδελφο Ματιέ, ο συνάδελφο ε, και ο κύριος Καζάκα επίσης από τους σοσιαλιστές είχε πάει πολλές φορές επί τόπου και δεν κατάφεραν να μάθουν τίποτα οπότε από ό,τι φαίνεται ακολουθούμε την αρχή πως ελπίζουμε να γίνουν τα πράγματα σωστά. Κοιτάξτε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν, δεν επαρκεί. Κάτι, κάτι θα πρέπει να γίνει ή να, να παρέμβουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο πρόεδρος. Υποθέτω πως Κομισιόν... έχετε κάποιο σχόλιο. Ναι, σύντομα. Ε, από την έκθεση Ματιέ. Ένα από τα αποτελέσματα της ήταν... πως ε, κάθε έξι μήνες ε, υπάρχει μια εκτίμηση της κατάστασης η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα και είναι στη διάθεσή σας βεβαίως συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, δίνει πληροφορίες για το τι κάνει εκεί πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πώς το κάνει. Δεν είναι τέλειο το σύστημα, το παραδέχομαι βεβαίω χρειάζεται βελτίωση, αλλά δεν είναι πως δεν ξέρουμε τίποτα, υπάρχουν πολλές πληροφορίες για αυτές μας. Μάλιστα, κύριο Γκάιρ. Θα ήθελα να σχολιάσω τις ε, ερωτήσεις που μου έγιναν. Ε, στο συγκεκριμένο ερώτημα του κ. Σόνεγκαρτ, όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να ελεγχθούν, να, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τα χρήματα των διεθνών δωρητών. Το αμερικανικό δίδαγμα είναι ότι χρειάζονται τεράστια ε, υποστήριξη για τη διαχείριση και αν υπάρξουν κάποιοι υπάλληλοι εκεί στη χώρα οι οποίοι πραγματικά εκπαιδεύσουν τους Αφγανούς υπαλλήλου και εισαγάγουν κάποια εργαλεία διαχείρισης, ε, κάποιες ε, αρχές που θα πρέπει να διαφυλάσσουν το σκόριο φθαλμού ε, ούτως ώστε η διοίκηση φτιάκ, οικοδομήσει μια διαχείριση η οποία να ανταποκρίνει τις δικές μας προδιαγραφές κάτι το οποίο δεν υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα. Εφόσον επιτευθεί κάτι τέτοιο, αυτή η εκμάθηση, τότε θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Αυτή είναι η αμερικανική εμπειρία. Ε, στο Υπουργείο Υγείας έκανα αυτή την προσπάθεια και αναφέρεται ότι πράγματι στο τέλος αυτής της προσπάθειας άρχισαν τα πράγματα στο Αφγανιστάν να λειτουργούν. Κάτω λοιπόν από αυτές τις προϋποθέσεις ε, υπάρχει μια ελπίδα εύρυθμης λειτουργίας και θεώρησα εγώ να πούμε ότι είναι σημαντικό να, εγγυηθεί, να, να εγγυηθούν οι Αφγανοί την ανεξαρτησία του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, ε, κάτι που επίσης δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Άρα η θέση μου είναι ε, ναι εφόσον και όχι όχι επειδή. Δηλαδή εφόσον εκπληρωθούν κάποιοι όροι ναι. Τώρα, τι γνωρίζουμε για την πραγματική κατάσταση στο Αφγανιστάν. Βεβαίω, εγώ έθεσα το ερώτημα στον εαυτό μου, θα πάω στο Αφγανιστάν ή όχι. Και αφού έγινε μια πρώτη συζήτηση με του συναδέλφου τη Επιτροπή, από όπου προέκυψε ότι η κατάσταση ασφαλεία ε, δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο στου υπαλλήλου τη Κομισιόν, τότε είπα ότι και εγώ δεν θα πάω. Ε, τα ερωτήματα λοιπόν ε, που τίθενται οι συνάδελφοι Βρυξέλλες ε, τα έλυσαν μέσω μιας βιντεοδιάσκεψης. Θεώρησα λοιπόν ότι η κατάσταση ασφαλείας δεν επιτρέπει να μεταβούμε εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε απολύτως καμία πληροφορία για το τι συμβαίνει εκεί. Και κατά τη διάρκεια της έρευνας ακούσαν πολύ γλαφυρές και ποικίλε ιστορίες σε σχέση με το τι γίνεται ε, με τους ε, δωρητές ε, οι οποίοι πάνε εκεί ε, και με ελικόπτερα και δημιουργούν ε, προσωρινά ένα, στείλουν ένα αυτοσχέδιο σχολείο. Τώρα το τι γίνεται αυτή τη στιγμή φύγουν δεν το ξέρουμε. Θα πρέπει να έχουμε κάποια αξιόπιστα δεδομένα εν σχέση με το πράγμα ευρωπαϊκά κονδύλια φτάνουν εκεί και πώς αξιοποιούνται. Ε, αυτό το κάνει κατά την άποψή μου η Κομισιόν, προσπαθεί να το κάνει ε, συνεργαζόμενη με τοπικές μη κυβερνητικέ ενώσεις ε, και όπου οι άνθρωποι αυτοί επειδή είναι Αφγανοί μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια, όχι απόλυτη ασφάλεια, αλλά μεγαλύτερη ασφάλεια μπορούν να πάρουν φωτογραφίες, να έχουν δορυφορικές λήψεις, να κινηθούν με GPS κλπ. Όλα αυτά γίνεται, Βεβαίως είναι μια... υπάρχει πόλεμος εκεί και δεν είναι δυνατό να κάνει κανείς μια, να κινηθεί όπως θα κινείται στο Μπάντεν wurttemberg επί παραδείγματι. Όσον αφορά την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, τα πράγματα είναι λίγο πιο ζωφερά από ό,τι πίστευα. Εγώ παραιτήθηκα από την προσπάθεια να καταλάβουμε ποιο κάνει τι. Γιατί ο επιμερισμό καθηκόνων μεταξύ των διαφόρων τμήματων τη ε, Επιτροπή μαζί με τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και η ορθέτηση των είναι τόσο μπερδεμένη και σχέση προς τις χώρες ε, μέλη. Οπότε παρατήθηκα από αυτή την προσπάθεια. Και άρα οι πληροφορίες που έχω είναι περιορισμένες η εντύπωσή μου είναι ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ κομισιών από την άλλη, τις αριστερότητες των χωρών μελών από την άλλη, ε, χρήζουν βελτιώσεων μεν, αλλά γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης. Είναι κάπως θολή, ε, αόριστη αυτή η διατύπωση βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά δείχνει κάποια ελπίδα η αοριστή αυτή. Η εντύπωσή μου είναι ότι από τότε που δουλεύει εκεί ο πρέσβης υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Το υπάρχει μια μικρή βελτίωση δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι ιδεώδη. Τώρα, μπορεί η βοήθεια του προπολογισμού να λύσει τα προβλήματα. Όχι βεβαίω είναι η απάντηση. Μπορεί να επιλύσει ορισμένα προβλήματα, το capacity building για παράδειγμα, και μέσω αυτού να προετοιμάσει κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να επιτελέσει το ίδιο το αφγανικό κράτος. Ε, Βεβαίως ε, αυτό δεν μπορεί να το κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ούτε οι ιδιώτες εταίροι, ούτε τα διαπιστεύματα μπορούν ε, να το πετύχουν. Γιατί αυτή τη στιγμή η αφγανική κυβέρνηση, η διοίκηση είναι όπως είναι, Άρα δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Άρα λοιπόν, ναι, δεν μπορούν να επιληθούν όλα τα προβλήματα μέσω αυτή τη ε, συνδρομή, αλλά μπορεί να βοηθήσουν τα χρήματα αυτά να λυθούν συγκεκριμένα προβλήματα που δεν λύνονται με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι κάλυψα όλα τα θέματα. Okay. Thank you. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Η προθεσμία για τροπολογίες είναι την ερχόμενη Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στις 12 η ώρα. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το 8 μελέτη για το ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, της υφιστάμενης νομοθεσίας ε, για έλεγχο αποτελεσματικότητας και ποιοτικό έλεγχο στις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων. Τι ρόλο μπορεί να παίξει ο έλεγχος απόδοσης. Ο Γιάννης Γκάιερ και εδώ πέρα είναι συγητής. Θέλετε τον λόγο πριν μιλήσουν οι ειδικοί. Όχι. είναι λοιπόν τον λόγο συντάκτης της μελέτης και υποθέτω πως μεταξύ σας έχετε ήδη συμφωνήσει ποιος θα μιλήσει πρώτος. Ο κύριος Μπλομάγερ. Θα σας παρουσιάσω σύντομα μία μελέτη που έγινε το πρώτο εξάμεινο του 2011. Λίγα λόγια για το περιεχόμενο αυτής της παρουσίασης. Θα πω κάποια πράγματα για τους κύριους στόχους της μελέτης και την μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα θα σας πω ποια ήταν τα ευρήματά μας και τις συστάσεις μας. Στόχος της μελέτης ε, ήταν να σας δώσει μια γενική εικόνα για τις διαφορετικές πτυχές ε, του ελέγχου διαρθρωτικών ταμείων και ταμείου συνοχής για να δείτε παραδείγματο χάρη ποιοι είναι οι διάφοροι φορείς του ελέγχου, ποια είναι η βασική τους προσέγγιση, ποιος είναι ο ρόλος ελέγχου απόδοσης σε σχέση με τον έλεγχο συμμόρφωσης, δηλαδή κοιτάμε το αποτέλεσμα που έχουν επιτύχει τα διαρθρωτικά ταμείου, ενώ ο έλεγχος συμμόρφωσης εξετάζει το εάν η δραστηριότητα υποστηριχθήσα ε, έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο. Η μελέτη επίσης έχει στόχο να σας δώσει μια ιδέα της ελεγκτικής προσπάθειας και το εύρος ε, του ελέγχου και ποιο είναι το ποσοστό των δαπανών και το τι καλύπτει και το κόστος βεβαίως. Και τέλος, ως ε, ένα γενικότερο στόχος να βρούμε πού μπορεί να βελτιωθεί η υπάρχουσα προσέγγιση για τον έλεγχο των διαρθρωτικών ταμείων. Τι κάναμε λοιπόν. Ήρθαμε σε επαφή με διάφορους ενδιαφερομένους σε διάφορα επίπεδα και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάναμε μια έρευνα μεταξύ 46 ελεγκτικών αρχών από 20 κράτη-μέλη και εξετάσαμε ειδικά διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα σε 8 ε, ε, κράτη-μέλη, Τσεχία, Ισπανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Αναζητούσαμε πρακτική εμπειρία για το πώς ε, οι φορείς αυτοί βλέπουν τις ελεγκτικές απαιτήσεις σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Οπότε, τα ευρήματά μας μία από τις πρώτες πτυχές που είδαμε είναι το ποιος εμπλέκεται και βεβαίως στόχος ήταν να μάθουμε κάποια πράγματα παραπάνω για τις πρακτικές εφαρμογές αυτού του οποίου λέμε μια προσέγγιση ενιαίου ελέγχου να μην γίνεται δηλαδή δύο φορές ο ίδιος έλεγχος. Γενικά η αντίδραση ήταν θετική, οι φορείς που εμπλέκονται ήταν οι ορισμένες ε, αρχές ελέγχου, κυρίως στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης και οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε θετικές ε, αντιδράσεις ειδικά όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας ε, που εισάγεται στο άρθρο 73 του ισχύοντος κανονισμού και επιτρέπει κατά βάση στους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βασιστούν στις ε, γνωμοδοτήσεις, τις ελεγκτικές που υποβάλλονται κάθε έτος από τις αρχές ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επιπλέον εξετάσαμε το ελεγκτικό έργο του ελεγκτικού συνεδρίου και από τα κράτη-μέλη, από τους, τους ελεγκτικούς φορείς, που είναι συγκεντρικό και σε ορισμένα κράτη-μέλη σε περιφερειακό επίπεδο. Η αντίδραση συνολικά ήταν θετική. Υπάρχει συντονισμός μεταξύ των αρχών για να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις, παραδείγματο χάρη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα από την Ισπανία. Παραδείγματο χάρη, οι Ισπανικές ελεγκτικές αρχές μας είπαν πως είναι ικανοποιημένε με τον τρόπο οργάνωσης ε, του συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν συμπίπτει ο δικός τους ο έλεγχος με τον έλεγχο των Ισπανικών αρχών. Επίσης, ε, μας ενημέρωσε για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Αν δείτε παραδείγματο χάρη τα ευρήματα των ελεκτικών αρχών, συνολικά γύρω στο 90% όσων απάντησαν, απάντησαν πολύ θετικά όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ των ελεκτικών αρχών της Ένωσης και των κρατών μελών. Ένα 70% είχε θετική άποψη όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις ε, όπου ίσως υπάρχει κάποιο, κάποιο περιθώριο βελτίωσης, π.χ. αν πριν από μία επίσκεψη μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών, αν ε, έχει γίνει ήδη παραδείγματο χάρη μία επίσκεψη από την Κομισιόν ή από το ελεγκτικό συνέδριο. Διαφορετικές λοιπόν οι εμπειρίες από τα 8 κράτη-μέλη και δεν ξέρω τώρα εάν ο κύριος Μπέρξ από τη Βορειορινανία Βεσφαλία θέλει να μας δώσει κάποιο παράδειγμα και να μας πει τι βρήκε συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, κάναμε δύο ξεχωριστές μελέτες για την κεντρική βοημία και την Βόρεια Βεσφαλία. Το θέμα είναι όπως διαπιστώσαμε στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, είναι πως η οργάνωση του ελέγχου είναι τέτοια ώστε τα, το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης ε, του Ταμείου Συνοχής οργανώνεται σε ένα δεύτερο επίπεδο από την ελεγκτική αρχή, αλλά βεβαίως υπάρχει και υψηλότερο επίπεδο συγχρηματοδότησης και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα του ελέγχου είναι το ελεγκτικό συνέδριο της ε, Ρινανίας Βασθαλίας και βεβαίως και το ελεγκτικό συνέδριο το ευρωπαϊκό που θα πρέπει να ελέγξουν ούτως ή άλλως αυτά τα προγράμματα και το πρόβλημα δεν είναι τόσο η αλληλεπικάλυψη η αναποτελεσματικό συντονισμός αλλά είναι η εντύπωση πως ε, το σύστημα είναι σχεδιασμένο όπως είναι και δεν υπάρχει τρόπος νομικός ε, να υπάρξει συντονισμός ε, μεταξύ όλων αυτών των αρχών των ελεγκτικών. Αντιθέτως μας είπαν πως εάν υπήρχε περισσότερος συντονισμός μεταξύ των περισσότερων των διαφορετικών ελεγκτικών αρχών θα υπήρχε ο κίνδυνος ε, απάτηση παρατυπιών και θα ήταν ακόμη ψηλότερος. Οπότε είναι εκπροθέσεως έτσι το σύστημα. Και ε, η περισσότερη αποτελεσματικότητα δεν θα επιτευχθεί μέσω του συντονισμού. Μάλιστα. Η μελέτη επίσης εξέτασε την ελεγκτική προσέγγιση, τι αναζητούν οι ελεγκτές, αν είναι η συμμόρφωση, αν είναι η απόδοση. Ξέρετε πως είχαμε συζητήσει αυτή την έννοια του έλεγχου απόδοσης. Συνολικά βρήκαμε πως το βάρος είναι σαφώς στην συμμόρφωση δηλαδή οτιδήποτε έχει γίνει να συμφωνεί με τις ε, απαιτήσει ε, τις ρυθμιστικές για τις δαπάνες αυτές. Και στην έρευνά μας λοιπόν και στις ε, ειδικέ περιπτώσεις ρωτήσαμε μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ απόδοσης και συμμόρφωσης. Όπως βλέπετε από τα νούμερα υπάρχει στήριξη για το υπάρχουν σύστημα, οι αρχές σε γενικές γραμμές θεώρησαν πως υπάρχει μια επαρκής ισορροπία μεταξύ των δύο, αν και βλέπετε πως ένα τέταρτο των όσων απάντησαν θεωρούσαν πως θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος έλεγχος της απόδοσης στα διαρθρωτικά ταμεία, πως δεν επαρκεί και στις περιπτώσεις που εξετάσαμε λεπτομερώς ε, είδαμε πως ε, Κάποιοι είχαν πρώτες εμπειρίες όσον αφορά την, ε, τον έλεγχο της αποδοτικότητας ε, και φαίνεται πως αυτό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ στα κράτη-μέλη, στα επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε, αλλά και συνολικά θεωρούν πως μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η πτυχή. Όμως υπάρχουν περιορισμοί και κάποιοι από αυτούς τους περιορισμούς ε, υπάρχουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο το ίδιο. Το ανέφερε ο κύριος Μπέργκς πως ε, το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο βεβαίως ρίχνει βάρος στον έλεγχο συμμόρφωσης και δεν αφήνει περιθώριο να εξτάσουμε την απόδοση. Κάτι άλλο το οποίο είπαν ε, διάφορα κράτη-μέλη είναι πως δεν υπάρχει εμπειρία και πόροι ε, περισσότερων ελέγχων απόδοσης. Μας είπαν πως δεν έχουμε αυτή την ε, εμπειρία, αυτό είναι κάτι που θα το δουν οι αξιολογητές, τα αποτελέσματα δηλαδή και τον ευρύτερο αντίκτυπο δεν το γνωρίζουμε το αντικείμενο. Όταν είδαμε λοιπόν κάποια κράτη-μέλη που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία με έλεγχο απόδοση, παραδείγματο χάρη στη Δανία, είδαμε πως ήταν ε, η διαδικασία μακροσκελής και χρειάζονταν χρόνος για να αποκτήσουν αυτή τη γνώση και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχαν αμφιβολίες αν αυτές οι ελεγκτικές διαδικασίες σχετικά με την απόδοση θα μπορούσαν να οδηγήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις και προσαρμογές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σαν παράδειγμα για την επιστροφή ε, ποσών που δεν θα έπρεπε να είχαν δοθεί. Δεν ξέρω για την τομέα της βιομηχανίας αν υπάρχει κάποια διαφορετική. Σχετικά με την ελεκτική διαδικασία μέσω της απόδοσης. Εξετάζεται η αποτελεσματικότητα φυσικά Μέχρι κάποιο σημείο όμως. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να δούμε είναι οι προθέσεις της παρέμβασης η οποία σχεδιάζεται και αν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί ή όχι. Αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο αξιολογώντας πλήρως τις αποδόσεις και τη λειτουργία του μηχανισμού ανάμεσα στην απόδοση από τη μία και την αποτελεσματικότητα από την άλλη. Προσπαθούμε να συγκρίνουμε τους δείκτες τους οποίους χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να πετύχουν τους στόχους τους αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται. Δίδεται επίσης αρκετά μεγάλο βάρος και στην αηφορία οι ελεγκτικές ε, υπηρεσίες ε, θα έλεγα είναι υποχρεωμένες να εξετάζουν και τα συστήματα λειτουργίας των συγκεκριμένων αρχών και δομών. Και εδώ τίθεται και το θέμα της συνέχισης λειτουργίας και παρουσίας των παρεμβάσεων αυτών στο μέλλον. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μία περιγραφή της παρούσης ελεγκτικής διαδικασίας, του εύρους της ελεγκτικής διαδικασίας, του όγκου της ελεγκτικής διαδικασίας και σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα πράγματι επαληθεύονται από τους ελεγκτές. Βλέπουμε ότι έχει υπάρξει αύξηση των δαπανών κατά πρώτον ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας των διαφορετικών ταμείων. Εδώ βλέπετε μια μικρή σύγκριση ουσιαστικά α, της περίοδου 2000-2006 και τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε από συγκεκριμένες μελέτες τις οποίες κάναμε είναι ότι τώρα ελέγχουμε όχι μόνο το 6% όπως τότε αλλά το 30% περίπου. Σαν παράδειγμα σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία και φτάνουμε στο 50 και 60% σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Βόρεια Βεσφαλία. Έχουμε λοιπόν πολύ περισσότερα στοιχεία και πολύ περισσότερα παραδείγματα προς έλεγχο από ό,τι είχαμε στο παρελθόν στη διάθεσή μας. Και ταυτόχρονα οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε τώρα μας επιτρέπουν να κάνουμε δειγματοληπτικές ελεγκτικές διαδικασίες πιο αποτελεσματικά. Αυτά βέβαια αυξάνουν και το κόστος της ελεκτικής διαδικασίας και αυτό το οποίο προσπαθεί η διαφάνεια να δείξει είναι από τη μία αποτελέσματα μιας τελευταίας μελέτης την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέγει ότι έχουν ελεχθεί 12 δις στα πλαίσια της διαχείρισής τους και το κόστος της ελεγκτικής διαδικασίας είναι περίπου το 8% συνολικά για τα ταμεία αυτά, τα διαφορετικά. Όταν βλέπετε τα διαφορετικά προγράμματα πιο κάτω στον πίνακα, βλέπετε όταν ένα εκατομμύριο κόστους ελεγκτικού ή μάλλον συνολικής δαπάνης 3.000 περίπου, 2.700 μάλλον δαπανώνται για την ελεγκτική διαδικασία. Και έχουμε και διαφορετικές κλίμακες βέβαια χώρα. Βλέπετε ότι στην Ολλανδία κοστίζει η ελεγκτική διαδικασία 12.800 εκατομμύριο, 17.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία λιγότερο, πολύ λιγότερο. Αυτά τα συζητήσαμε και με τον κύριο Γκάγερ για να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία και όχι μόνο αριθμούς. Αλλά νομίζω ότι οι αριθμοί δεν είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστοι, είναι αλήθεια. όλα γίνονται σε μια βάση θα έλεγα ελεγμένη ένα αλλά ταυτόχρονα εμπειρική σε αυτή τη φάση. Έχουμε ξεκινήσει, θυμίζω, σχετικά πρόσφατα και δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για τον τρόπο ερμηνείας των στοιχείων αυτών. Και νομίζω λοιπόν ότι τα στοιχεία που έχουμε για το 2007 σαν παράδειγμα που έχουμε χρησιμοποιήσει δεν είναι ιδιαίτερα πλήρη. Αυτό θέτει ένα θέμα. Η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι δικαιολογημένη και πρέπει να συνοδεύεται και από τις παραδοσιακές ελεκτικές διαδικασίες. Εδώ θα πρέπει να δούμε πραγματικά το κόστος της ελεκτικής διαδικασίας σε σχέση με την βελτίωση των αποτελεσμάτων. Αν δείτε σαν παράδειγμα για το Περιφερειακό Ταμείο τα στοιχεία, αλλά και για άλλα ταμεία επίσης όπως το Ταμείο Συνοχής, Βλέπετε ότι έχουν δαπανηθεί, έχουν διορθωθεί ποσά, έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί ποσά που φτάνουν περίπου τα 6,7 δις. 0,6 δις κατέτος χοντρικά τα τελευταία 10 χρόνια. Και αυτό μπορείτε να το συγκρίνετε αν θέλετε και με το κόστος της ελεγκτικής διαδικασίας. Το θέμα δεν είναι να συγκρίνουμε τα ποσά από τη μία και το κόστος ελέγχου από την άλλη. Το θέμα είναι για να καταλήξει κανείς σε καλά συμπεράσματα πρέπει να δει ποιε είναι οι ποιοτικέ βελτιώσεις, τα ποιοτικά πλεονεκτήματα τα οποία σημειώνονται. Και αυτό έχει γίνει από τις ανώτατες ελεγκτικές αρχές, μια ομάδα ανώτατων ελεγκτικών αρχών. Τα αποτελέσματα αυτών των αρχών δεν είναι απόλυτα δημοσιευμένα ακόμα. Είδαμε πάρα πολλά στοιχεία πάντως για την Πολωνία και εκεί υπογραμμίζεται η ποιοτική βελτίωση. Βελτίωση ποιονική που οδηγεί απλά στην καλύτερη διαχείριση των προγραμμάτων στο μέλλον. Γιατί η ελεκτική διαδικασία αποδεικνύει ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι, πιο αποτελεσματικοί τρόποι για τη διαχείριση των προγραμμάτων και γι' αυτό πρέπει να γίνουν αλλαγές στο μέλλον. Now seem, uh, there seems to be a problem with the um, uh, presentation. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με την παρουσίασή μου από ό,τι φαίνεται. I think we continue without these slides. Um, just one second. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε χωρίς τις διαφάνειες. Ωραία λοιπόν, έμειναν δύο διαφάνειες, άρα δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά παρόλα αυτά θα ήταν καλό να τις βρίσκαμε γιατί έχουμε κάτι γράφικς τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ωραία λοιπόν, ε, ήταν ακόμα δύο διαφάνειες. Έστω θα τις αφήσουμε. Έχετε τα έγγραφα. Ζητήσαμε ε, να μας πούν οι ελεγκτικές ε, αρχές ε, κατά πόσο υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά την ωφέλεια αναγνώρισης κάποιων ατασταλιών σε σχέση με το κόστος. Πολλοί θεωρούν ότι ναι. 80% ε, μας είπαν ότι πράγματι ε, έχει νόημα κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. 12% των αποκρινόμενων της μελέτη λένε ότι θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να ενισχυθεί αυτή η διαδικασία ελέγχου. Κάποια τελικά λοιπόν σημεία. Οι συστάσεις. Κάτι το οποίο προέκυψε εντόνως από όλες τις συζητήσεις είναι ότι χρειάζεται να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά σε μέτρα πλούστευσης καθώς θα γνωρίζετε υπάρχει μια υποεξέλιξη μελέτη η οποία εξετάζει ειδικά ορισμένα από αυτά τα μέτρα πλούστευσης και πολλοί από τους ελεγκτές το εξέφασαν με τις εξής ώρες. Τα περισσότερα πράγματα τα οποία ε, αντιμετωπίζουμε είναι θέματα επιλεξιμότητας τα οποία γύρει το εξαιρετικά πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσπάθεια να υπάρξει μια πλούστευση χωρίς ε, βεβαίως να γίνουν και πραγματικές επαναστάσεις ε, όχι να ανατροπεί όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο και να αλλάξει εκβάθρων. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να βελτιωθεί και να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιστροπής και χωρών μελών. Ενισχύοντας λοιπόν αυτή την ελεγκτική προσέγγιση βήμα προς βήμα. Ε, βρήκαμε μεγάλη υποστήριξη λοιπόν και γι' αυτό σας συστήνουμε την ε, περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ε, διαδικασίας ελέγχου ούτως ώστε να αποφευθούν κάποιες ε, επικαλύψεις να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπιστευτεί τη γνωμοδότηση των ελεγκτικών αρχών και πιστεύουμε επίσης ότι η ελεγκτική προσπάθεια θα πρέπει να σχετιστεί περισσότερο με το μέγεθο των προγραμμάτων, για τι των προγραμμάτων, να επικεντρωθεί δηλαδή σε μεγαλύτερα προγράμματα. Επίση, η ελεγκτική προσπάθεια θα πρέπει να αξιολογηθεί περισσότερο όσον αφορά την επίδοση ενό ε, λειτουργικού, την απόδοση ενό λειτουργικού προγράμματο. Αν έχετε ένα λειτουργικό πρόγραμμα το οποίο για πολλά χρόνια κατά την άποψη του ελεγκτού υπήρξε θετικό και δεν έχουν αναγνωριστεί καθόλου προβλήματα, τότε ενδεχομένω μπορείτε να μειώσετε την προσοχή που προσδίδεται σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να εστιάσετε κάπου αλλού. Και τέλος βρήκαμε πολύ ισχυρή υποστήριξη και αυτή είναι η τελευταία σύσταση την οποία κάνουμε στην έκθεσή μας για μια περαιτέρω ανάπτυξη στοιχείων ελέγχου πίδωσης. Πολλές χώρες μέλη έδειξαν σχετικά ενδιαφέρον. Και μπορεί να συνεχίσει λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Όχι, πραγματικά οι τελευταίες δύο διαφάνειες μοιάζει να έχουν εξαφανιστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία και πάλι θα αναλάβω την Προεδρία. Ε, χρειάστηκε να εγκαταλείψω λίγο την αίθουσα. Δεν ε, άκουσα λοιπόν την παρουσίαση. Συγγνώμη, ε, θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Ε, ο πρόεδρος και η γραμματεία εξαφανίστηκαν. Γενς. Ναι. Ε, θα τα καταφέρουμε και χωρίς γραμματεία και χωρίς πρόεδρο. Μην ανησυχείτε. Έχω δύο σημεία, τα οποία αφορούν και την εργασία της Επιτροπής μας. Πρώτον, θα πρέπει να σκεφτούμε, πιστεύω, το πόσο μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάπως τα καθήκοντά μας, ε, για τις, ε, τους στόχους μάλλον για αυτές τις μελέτες και τα δικά μας καθήκοντα. Δηλαδή παράγουμε πάρα πολλές ιδέες, ακούγονται θαυμάσια και τελικά υπάρχει, υπάρχουν περισσότερες ιδέες παρά ικανότητε στο τέλος, δυνατότητες. Ε, και ε, προσπαθούμε να συνενώσουμε κάποιες ε, προβληματικές, ε, κάτι το οποίο δεν επιτυγχάνεται πάντοτε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε συνολικά να διευκολύνουμε το βίο των εμπειρογνωμόνων μας εάν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επί ενός μηχανισμού για το πώς μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε απολύτως τους σκοπούς μιας έρευνας, μιας μελέτης. γιατί είναι αρκετά ακαθόριστη, αόριστη αυτή η σκοπή. Ε, και καμιά φορά θεωρώ αν είχαν γίνει δύο μελέτες, ίσως τα αποτελέσματα θα ήταν πιο ξεκάθαρα, αντί για μία επί παραδείγματι. Ε, στον κύκλο αυτό ε, συστήσαμε πολύ και με το ελεγκτικό συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σε σχέση με τις αναλύσεις των αποτελεσμάτων. Και αν το συγκρίνω με αυτό με τα αποτελέσματα των Πλήμαρ και Σάντς, και με αυτό που θα μπορούσαμε να προσμετρήσουμε κάτω από τις σημερινές συνθήκες νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε στη διάθεσή μας το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν έχουμε τη βάση της συνθήκης βάση της οποίας θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο Υπάρχουν βεβαίως οι προσδοκίες σε ορισμένες χώρες μέλη να γίνει κάτι τέτοιο και ίσως θα έπρεπε να εθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να το κάνουν ήδη, να απτύξουν μάλλον κάποιες ιδέες σε σχέση με το πώς θα πρέπει να συνεχίσουμε και με ευχαρίστησή μου θα συμμετάσχω στην περαιτέρω, στον περαιτέρω διάλογο με το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε τι δικέ μα προσπάθειε σε άλλου τομεί, γιατί χωρί νομική βάση, χωρί μια επιστική δέσμη παραμέτρων για το πώ θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό ο έλεγχο επίδοση, το performance audit, χωρίς την ε, προθυμία των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν, ε, νομίζω ότι όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε επακριβώς ποια είναι τα επόμενα βήματα. Εμένα με εντυπωσίασε, με εντυπωσίασαν διαφορετικά κόστη Ε, νομίζω ότι είναι κάπως ολισθηρό το έδαφος, αν κατάλαβα καλά από τον Μπλομάιρ. Γιατί τα αίτια της ε, παραγωγής κόστους είναι ασαφή. Εάν ε, δούμε το κόστος που διαφοροποιείται από το παράγοντα 10, ε, ίσως ορισμένοι τα κάνουν τα πράγματα τελώς λάθος, οι άλλοι τα κάνουν σωστά. Και πάντοτε ερχόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι οι εταίροι μας ε, παραπονούνται για αυτή την πληθώρα και πυκνότητα ρυθμιστικών κανόνων. Γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να ακούσουμε τη δική τους άποψη. Τι θεωρούν αυτοί οι ίδιοι ότι θα πρέπει να γίνει. Ε, και ποιο είναι ακριβώς το κόστος το οποίο θα πραγματικά θα πρέπει να υποκινήσει ακριβώς ένα, μια ρυθμιστική προσπάθεια. Η... Γερμανία συνήθω παίρνει εδώ την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά την ερμηνεία των ρυθμιστικών κανόνων, ούτε ώστε να δείξει ότι οι κανόνες αυτοί είναι πολύ πιο σημαντικοί από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και ίσως κάνουμε κάτι αντίστοιχο και στο θέμα αυτό των ελέγχων επίδοσης, των audits δεν ξέρω ή αλλιώς προσπαθούμε με το κόστος αυτό να έχουμε ένα ε, ε, να έχουμε κάποια καλύτερα εργαλεία αξιολόγησης των σφαλμάτων αλλά νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι πρόκειται για μια ιδέα που αρχικά ήταν αληθής ε, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι από τη μια μεριά είναι αυτό το κόστος, από την άλλη να μην είναι ξεκάθαρη η σχέση κόστους ωφέλειας. Το ερώτημα σχέση με την περαιτέρω απλούστευση, χωρίς όμως μια επανάσταση αν θέλετε κύριε Μπλομάιερ, μου δίνει λαβή σε κάποιες σκέψεις, σε κάποιες ερωτήσεις προς την κατεύθυνσή σας. Είναι δύσκολο κατά πάσα πιθανότητα να απαντηθεί, αλλά η ερώτηση πού θα μπορούσε να γίνει μια απλούστευση. Πού θεωρούν οι ενδιαφερόμενοι ότι θα πρέπει να γίνει απλούστευση και πού θα ξεκινούσε μια πραγματική επανάσταση όπως την αποκαλέσατε. Αυτό σαν επισήμανση για μια ακριβέστερη περιγραφή εκ μέρου σας. Ευχαριστώ. Προτείνω να ακούσουμε τα ερωτήματα κατόπιν των κύριων Χατζημαρκάκη Γκάσλε. Ναι, συμφωνώ απολύτως όσον αφορά αυτή την απλοποίηση την οποία αναφέρατε. Ε, μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν γίνεται αυτή η απλούστευση, γιατί αυτή η απέτηση του Κοινοβουλίου της Επιτροπής Θεμάτων να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες σε όλα τα ταμεία, γιατί δεν ε, ακολουθείτε και τι αποτέλεσμα έχει αυτό στο κόστος. Δηλαδή αυτή η διαφορά στο κόστος είναι φοβερή. Εάν ε, η ερώτηση είναι εάν ε, η απλοποίηση θα επέφερε και μείωση στο κόστος. Όσον αφορά τώρα τον έλεγχο απόδοσης, αυτό είναι το δεύτερο μου ερώτημα, στην ε, τελευταία έκθεση απαλλαγής της Κομισιόν είπαμε ξεκάθαρα πως με τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει καθήκον της Κομισιόν να κάνει έλεγχο απόδοσης. Και Είπαμε πως θα έχουμε μια συζήτηση κάθε χρόνο με το ελεγκτικό συνέδριο, δηλαδή να μην ε, κοιτάμε μόνο την ομόταλα και το τι αποτέλεσμα έχουμε. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει ένας τέτοιος έλεγχος απόδοσης, γιατί συγκεκριμένα δεν έχουμε κάτι ακόμα από την Κομισιόν. Ξέρουμε πώς θα έρθει κάτι. Τι ε, θα κάνατε εσείς ως έλεγχο απόδοσης, με ποια κριτήρια. Ευχαριστώ, Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Θα ε, έχω κάποιες ερωτήσεις ε, κατανόησης που ίσως να οφείλονται στο ότι συζητήσαμε τόσα πολλά θέματα, αλλά θα ήθελα να πω πως ε, όσον αφορά την κατεύθυνση της μελέτης θα πρέπει και εσείς να να κινητοποιηθείτε ε, και αυτός ο οποίος ανέθεσε την ε, μελέτη. Δηλαδή, κύριε Μπλόμαρ, πείτε μας με δύο λόγια πού πρέπει να εργαστούμε, τι πρέπει να κάνουμε. Δεύτερον, κάτι το οποίο με εντυπωσίασε ήταν οι διαφορές στο κόστος του ελέγχου. Μιλήσατε για μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην ε, μελέτη αυτή βασίστηκαν διάφορες ε, υποθέσεις και από ό,τι φαίνεται η μελέτη αυτή έχει τις χαμηλότερες εκτιμήσεις από όλες τις άλλες για το κόστος. Οπότε το ερώτημα είναι πώς γνωρίζουμε ποιο είναι το πραγματικό ύψος του κόστου του ελέγχου. Οπότε θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε πού μπορούμε να βασιστούμε όσον αφορά ακριβώς αυτή την αξιοπιστία του κόστους του ελέγχου. Ο κύριος Σταυρακάκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σχολιάσω ορισμένα από τα σημεία της μελέτης. Πρώτον, στη μελέτη σημειώνεται ότι η αυξανόμενη προσπάθεια ελέγχου έχει οδηγήσει σε ανάλογη αύξηση του κόστους ελέγχου όπως έχει επανειλημμένα υποστηρίξει τόσο η Επιτροπή περιφερειακή Ανάπτυξης όσο και αυτή εδώ η Επιτροπή οι έλεγχοι που σχετίζονται με τα διαφορετικά ταμεία και με το Ταμείο Συνοχής δεν θα πρέπει να δημιουργούν μια δυσανάλογη επιβάρηση τόσο για τους ελεκτές όσο και για τους ελεγχόμενους. Υποστηρίζουμε τις αρχές της αναλογικότητας και της προσέγγισης ενιαίου ελέγχου, single approach, φυσικά να παραβιάζεται η αρχή ότι το κάθε ευρώ του Ευρωπαίου φορολογούμενου πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά. Δεύτερον, ένα από τα πιο ενισχυτικά συμπεράσματα που προκύπτει από την εξέταση των περιπτώσεων στα διάφορα κράτη-μέλη είναι ότι το πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχή αναγνωρίζεται ω μία από τι βασικέ αιτίε που προκαλούν παρατυπίε. Δεν μπορώ κι εγώ παρά να υπογραμμίσω την ανάγκη για απλοποίηση κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι αν και η μελέτη παρέχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, δεν προβαίνει σε βάθος ανάλυση. Επιπλέον, δεν προσφέρει ουσιαστικέ προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου των διαφορετικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Er eh, Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει το λόγο. Όχι. Οπότε έχετε εσείς τον λόγο. Κάποια γενικά σχόλια για τις μελέτες τις οποίες κάναμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Και πάντα ανησυχούμε όταν βλέπουμε εμείς τους όρους να περιγράφουν τη δουλειά μας και οι οποίοι είναι πάρα πολύ γενικόλογοι και μερικές φορές ε, δεν τίθενται αν θέλετε τα σωστά ερωτήματα και δεν συναρτώνται μεταξύ τους. Και τώρα είχα κάποιες ανησυχίες και λόγω χρόνου και αυτό το οποίο προτείναμε εμείς σαν ομάδα είναι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα θέματα. Ίσως στο μέλλον θα ήταν καλύτερο να έχουμε περισσότερες ενδιάμεσες συναντήσεις έτσι ώστε να έχουμε σωστούς στόχους τουλάχιστον ιδιαίτερα σε σχέση με την μελέτη για την απλούστευση των διοικητικών μέσων μέτρων, προτείνεται να έχουμε μια ειδική συνάντηση στα πλαίσια της οποίας θα μπορέσουμε να εξετάσουμε λεπτομερέστερα το στόχο αυτό. Λοιπόν, αυτό το οποίο προσπαθούμε λοιπόν είναι να σας δώσουμε ένα χρήσιμο σε εισαγωγικά άρωμα του τι κάνουμε και ποιες είναι οι πρακτικές οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα κράτη-μέλη, να σας δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα λειτουργικών προγραμμάτων, να εξετάζουμε τα προγράμματα αυτά και να επιλέγουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβετε καλύτερα. Σχετικά με το κόστος, για αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα το εξετάζουμε φυσικά στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία σαν παράδειγμα. Συγκρίναμε το κόστος το ελεγκτικό του προγράμματος αυτού. Νομίζω λοιπόν ότι ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση το κόστος σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνάει ανεκτά ποσοστά. βλέπετε πως ε, μια συγκεκριμένη χώρα βεβαίω έχει το υψηλότερο ποσοστό ελέγχου, οπότε θα είναι θαυμάσια η έλεγχη. Τέλο, θα φτάσουμε την έλεγχη. Λοιπόν, για τον έλεγχο της, ε, για τη μελέτη τη Κομισιόν, πράγματι είναι ένα πολύ καλό έγγραφο που κοιτάει διάφορε πτυχέ, αλλά αναγνωρίζει πω ίσω να έχει συνταχθεί κάπω νωρί όσον αφορά τον έλεγχο. Γιατί όταν κοίταζε το κόστο τη διαχείριση των ε, προγραμμάτων, υπάρχουν πολλές εξηγήσει για το πρόγραμμα και για το πώς ξεκινάνε τα προγράμματα, αλλά όχι για τον έλεγχο. Γιατί, Γιατί ο έλεγχος γίνεται στο τέλος όταν έχουν γίνει οι δαπάνες. Οπότε η μελέτη αυτή αναγνωρίζει η ίδια πως κάποια από τα στοιχεία αυτά είναι εκτιμήσεις που θα πρέπει βεβαίως μετά να επαληθευτούν. Όσον αφορά λοιπόν την επαλήθευση, μπορούμε απλά να σας δώσουμε παραδείγματα από αυτές τις 8 ή 9 περιπτώσεις για τις οποίες έχουμε δεδομένα. Σε κάποιε περιπτώσει δεν υπάρχουν δεδομένα. Στην Ισπανία, παραδείγματο χάρη, είχαμε μια συνάντηση με την ελεγκτική αρχή, την κεντρική, και λάβαμε πολλέ πληροφορίε, αλλά είχαμε μηδενικέ πληροφορίε για το κόστο του ελέγχου και πιθανώ ε, ανάλογη θα είναι η κατάσταση σε πολλέ ε, χώρε. Τώρα, στι χώρε εκείνε τι οποίε έγινε η προσπάθεια, και η προσπάθεια έγινε στο πλαίσιο μελετών ε, δύσκολων, π.χ. στην Ολλανδία ακολούθησαν διαφορετικές μεθόδους και κατέληξαν και σε διαφορετικά αποτελέσματα. Οπότε ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζει κανείς καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα μεταξύ 12.000 και 30.000 ευρώ ανά ε, εκατομμύριο ευρώ ελεχθέντος ποσού. Οπότε δεν υπάρχει κάποια στη βαρύ εμπειρική βάση από τα έγγραφα τα οποία είδαμε εμείς για το κόστος του ελέγχου. Επίσης, και αυτό επίσης είναι προφανώς ε, κοινή λογική, το κόστος ε, του ελεγκτή, της ώρας εργασίας του ελεγκτή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στη Φιλανδία δηλαδή υποθέτω πως είναι υψηλότερο το κόστος από ό,τι σε κάποια άλλα κράτη-μέλη στο Νότο ή στα νέα κράτη-μέλη. Και αυτό συνυπολογίζεται. Επίσης, ε, για την Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Να, ε, να σας πω γενικά. Για να ξεκαθαρίσω λίγο αυτό το πρόβλημα με την διακύμανση του κόστους. Νομίζω πως μέρος της διακύμανσης αυτής εξηγείται ε, με τις διαφορετικές μεθόδους δειγματοληψίας. Π.χ. εφαρμόζουν δειγματοληψία νομισματική μονάδα όπω λένε στην ε, Ρινανία Βεσφαλία και αυτό σημαίνει πω καλύπτουν μεγάλε παρεμβάσει και οι μικρότερε δεν καλύπτονται τόσο. Οπότε εδώ πέρα έχουμε εφαρμόζουμε κατ' ουσίαν την μέθοδο της, ε, του επίπεδου σημαντικότητας. Εάν έχουμε δηλαδή ένα επιχειρηματικό κεφάλαιο και το ελέγχουμε είναι φτηνό ανα, αναμονάδα εξορισμού γιατί βεβαίως είναι μεγάλα τα ποσά, μεγάλες παρεμβάσεις και το ελέγχουμε μία φορά και έχει είναι πολύ μεγάλο το έργο οπότε τα μεγάλα αυτά έργα τα οποία ελέγχονται μειώνουν το μέσο κόστος του ελέγχου και αυτή η διακύμανση βεβαίως ε, οφείλεται και σε διαφορετική ερμηνεία βεβαίως το τι εννοούμε κάθε φορά, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στις διαφορετικές μεθόδους δειγματοληψίας. Ένα άλλο σημείο που αναφέρθηκε για το γιατί δεν υπάρχει επανάσταση Παρακολουθούμε στενά τις συζητήσεις στα κράτη-μέλη και σε ό,τι βλέπουμε μεταξύ κομισιών και κρατών μελών για την προετοιμασία του νέου πλαισίου που ε, προσεχώς βεβαίως θα έρθει υπό μορφή πρότασης. Η εντύπωσή μας από τις ε, διαχειριστικές αρχές τι οποίες γνωρίζουμε στη χώρα μας και τα έγγραφα τα οποία βλέπουμε η στήριξή τους για απλοποίηση, για βελτίωση του συστήματος, αλλά όχι για ολοκληρωτική ε, αλλαγή του, είναι αυτό το οποίο προτιμούν. Γιατί, γιατί οι ελεγκτικές αρχές υποφέρουν από το πολύπλοκο αυτό πλαίσιο, γιατί έχουν περισσότερη δουλειά και αυτό εξηγεί βεβαίως ε, και την ε, απροθυμία τους για μια επανάσταση και ολοκληρωτική αλλαγή γιατί βεβαίως έχουν επενδύσει στο να μάθουν και να στήσουν αυτό το σύστημα το οποίο λειτουργεί τώρα οπότε λένε σας παρακαλώ μην το αλλάξετε εκ βάθρων. γιατί θα έχουμε πάλι νέο κόστος θα πρέπει να το ξαναμάθουμε και θα χάσουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια για να μάθουμε το νέο σύστημα και να ερμηνεύσουμε σωστά το νέο σύστημα. Οπότε υπάρχει στήριξη για μικρές σταδιακές αλλαγές μέτρα απλοποίησης. Υπάρχει γενικά πάρα πολύ στήριξη όσον αφορά τις ε, απλοποιημένες ε, ε, επιλογές κόστους που υπάρχουν. Επίσης υπήρχε το ερώτημα αυτό απλοποίηση τη ελεγκτική προσέγγιση. Μα ρώτησαν γιατί δεν συζητάτε περισσότερο όταν προετοιμάσετε το δείγμα σα ω ελεγκτική αρχή, γιατί δεν κοιτάτε τι έχουν ελέγξει οι άλλοι σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο και αναλόγω να το αλλάξετε. Εδώ πέρα υπάρχει ένα νομικό ζήτημα α, περί ανεξαρτησίας των διαφορετικών θεσμικών οργάνων που κατ' ουσίαν δεν του επιτρέπει να λάβουν υπόψη α, τέτοια πράγματα και να έχουν έτσι κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Δηλαδή τους επιτρέπει σε γενικές γραμμές, αλλά όχι να αλλάξουν ε, το πώς κάνουν ε, τη δειγματοληψία. Επίσης, ο κύριος Σταυρακάκης ανέφερε κάτι σωστό, δηλαδή το να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Αυτό είναι το βασικό εδώ πέρα. Και πράγματι, ε, ειδικά σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία αποδίδουν καλά, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε πράγματι αξίζουν ε, πλέον ε, να τους εμπιστευτούμε. Έχουν αποδώσει καλά υψηρά ετών. Δεν χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε συνέχεια σε αυτούς. Και πράγματι ως ένα βαθμό αυτό συμβαίνει ήδη, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης νομίζω είναι παρούσα στην αίθουσα. Τους βλέπω εκεί πέρα, ίσως μπορούν να σχολιάσουν για το συγκεκριμένο αυτό θέμα της αναλογικότητας. Goed. Ehm, είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση. Όλοι και ο εισηγητής. Ναι. Ωραία. Οπότε τελειώνουμε με αυτό το θέμα, εκτός εάν... Α, η Κομισιόν θέλει τον λόγο. Βεβαίως. Ε, με συγχωρείτε που δεν ε, κοιτάω προς τα εκεί. Λοιπόν, ε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Από την πλευρά της Επιτροπής θα ήθελα να πω κάποια πράγματα ε, υπό το πρίσμα της μελέτης, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μας, ιδιαίτερος ε, γιατί δεν συμμετείχαμε στη μελέτη. Και είδαμε ότι έχει διαβούλευση με πολλούς ενδιαφερόμενους στις ε, χώρες μέλη. Η, με εμά δεν έγιναν διαβουλεύσεις, ε, και ε, λυπόμαστε λίγο γι' αυτό. Γι' αυτό ε, χαιρόμαστε που μπορούμε να δώσουμε την άποψή μας σήμερα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα και να διαπιστώσουμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αντανακλούν τις ε, βελτιώσεις που έγιναν στα προγράμματα τόσο σε ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς όρους. Ε, πράγματι αναφέρθηκε ε, η αύξηση του κόστους του ελέγχου, αλλά υπάρχει και μια βελτίωση των αποτελεσμάτων. Από την πλευρά της Επιτροπής, αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μας είναι να γίνουν πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι ως προς το κόστος. Ε, και υπάρχει μια κάλυψη για την περίοδο 2007 2010 ε, υπάρχει μια ενημέρωση εκ μέρους των χωρών μελών και εκ μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου. Έτσι μπορούμε, νομίζω ότι πράγματι μπορούμε να εμπιστευτούμε περισσότερο τις ελεγκτικές ε, αρχές. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με θέματα που έθιξαν κάποιοι βουλευτές σήμερα εδώ και σε σχέση με κάποια στοιχεία της ε, έκθεσης. Είναι προφανές ότι οι χώρες μέλη θέλουν να έχουν ένα πιο σταθερό και ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο και η καλύτερη απλούστευση ίσως είναι να μην γίνουν ε, αλλαγές. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να γίνει κάποια απλούστευση ε, όσον αφορά το κόστος. Επίσης, όσον αφορά τα σφάλματα, όταν ε, κάναμε μια ανάλυση σφαλμάτων στη πολιτική της συνοχής, είδαμε ότι πολλά που θα αφορούν σφάλματα επιλεξιμότητας, ε, για παράδειγμα όσον αφορά τις δημόσιες ε, προμήθειες. Ε, αυτή είναι μια σημαντική πρόκληση τόσο για τις χώρες μέλη όσο και για την Κομισιόν τους ώστε να προστεύσουν ακόμα περισσότερο τους κανόνες τους. Όπως ξέρετε ότι ήδη έχουν διατυπωθεί οι κανόνες επιλεξιμότητας στο επίπεδο των χωρών μελών. Άρα υπάρχει μια δυνατότητα εκ μέρους των χωρών μελών να το κάνουν και τους συστήνουμε πραγματικά να προχωρήσουν σε μια απλούστευση ούτω ώστε να μην είναι ιδιαίτερω πολύπλοκοι οι κανόνε επιλεξιμότητα. Συνεργαζόμαστε με τι χώρε μέλη σε προληπτικό επίπεδο, επίση ε, παρεμβαίνοντα, ε, κάνοντα κάποιε διορθώσει και η βασική ιδέα είναι να έχουμε τη σωστή ισορροπία. Και μιλάω για ποσοστά σφαλμάτων, γιατί πάντοτε πρέπει να το κάνω ε, πριν φτάσουμε στους ελέγχους επίδοσης. Για το τελευταίο πρόγραμμα είχαν περισσότερα ποσοστά σφάλματο όσον αφορά την πολιτική συνοχή και γι' αυτό δεν ήταν δυνατόν για μα την Κομισιόν να έχουμε πολλούς πόρου για τον έλεγχο επίδοση. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε το 2011, ξεκινήσαμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα στον αφορά τη στρατηγική ελέγχου ε, στην περιφερειακή πολιτική και αυτό γίνεται τόσο στο επίπεδο του ελέγχου των προγραμμάτων, της οικονομικής διαχείρισης και κοιτάμε επίσης και νέα θέματα που μπορούν να είναι το αντικείμενο του ελέγχου επίδοσης, απόδοσης. Ε, αυτό πηγαίνει στην κατεύθυνση του, ε, της του νέου ρυθμιστικού πλαισίου προτίθεται να εκπονήσει η Κομισιόν. Θέλουμε να έχουμε μια εμπειρογνωμοσύνη ε, βάσει της εμπειρία του τελευταίου έτους, ούτε ώστε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την βελτίωση του ελέγχου απόδοσης. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να αντιδράσει σε αυτό. Όχι. Ωραία, λοιπόν σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συμβούλους για αυτά τα οποία μας παρουσίασαν. Οπωσδήποτε να τα λάβουμε υπόψη. Και τελειώνουμε με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το ένατο Έχουμε μία έκθεση για την επίσκεψή μας στο Κοσφοπέδιο και κοιτάω εδώ πέρα τον κύριο Σταυρακάκη στην ε, πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και ήταν έντονη η επίσκεψη πρέπει να πω είχα την τιμή να ηγηθώ αυτής της επίσκεψης και ήταν ιδιαίτερη υπό την έννοια πως η ισορροπία δεν υπήρχε στην παρουσία των πολιτικών ομάδων, δηλαδή δεν υπήρχε κανείς από το ΕΛΚ και τους φιλελεύθερους, αλλά πρέπει να πω πως ήταν ενδιαφέρουσα επίσκεψη, έντονη και συναρπαστική κάποιες στιγμές, υπό την έννοια πως κάποιες στιγμές ε, μας άφησαν ε, σε λάθος ε, μεριά των συνόρων και αναζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολόκληρη την αντιπροσωπεία και πανικοβλήθηκε. Αλλά βεβαίως ως ε, βουλευτές πήραμε μετά ένα λεωφορείο της γραμμής ε, και περάσαμε στην πρώην Ιεκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκεί που έπρεπε να βρεθούμε. Η έκθεση νομίζω ότι την έχετε λάβει ήδη. Για όσους ε, δεν ήταν παρόντες, ε, νομίζω πως ε, ήταν μια καλή ευκαιρία να ενημερωθούμε και θα ενημερωθείτε και εσείς ούτως ή άλλως από την έκθεση αυτή. Τώρα, Κυρίως ασχοληθήκαμε με το Κοσφοπέδιο, η επίσκεψη στη Φιρόμ ήταν ε, ιδιαίτερη γιατί είχαν γίνει μόλις οι βουλευτικές εκλογές ε, και σχηματίζονταν η κυβέρνηση, η πολιτική κατάσταση ήταν κάπως πιο δύσκολη και περιοριστήκαμε στο τι ε, σε κάποια πολύ συγκεκριμένα έργα που γίνεται στην πρώην Κοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και είχαμε μια πολύ αναλυτική ενημέρωση με τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έκθεση διαπιστώνω πως αυτό το οποίο ε, με το οποίο συμφωνούν και οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν παρόντες ε, κάποιες ε, συστάσεις λέει τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να σας τα διαβάσω όλα αυτά. Υποθέτω πως ε, θα έχετε ρίξει μια ματιά. Ο βασικός τόνος της επίσκεψής μας στο Κοσφοπέδιο είναι βεβαίως ε, πως ε, είναι σημαντική η προσπάθεια η οποία γίνεται. Βασική παρατήρηση είναι πως είμαστε παρόντες ως Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά θεσμικά όργανα, με διάφορους τρόπους παρέμβασης και το ερώτημα είναι εάν υπάρχει μια γενική εποπτεία, εάν υπάρχει μια αποτελεσματική διαχείριση ε, όλων όσων γίνονται, εάν ε, υπάρχει επίσης αναφορά στην Επιτροπή μας, ε, εάν θα πρέπει να ζητήσουμε ίσως περισσότερες πληροφορίες. Επίσης παρατηρήσαμε πως όσον αφορά την παρακολούθηση η οποία γίνεται πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες η ε, Όλαφ είχε κάνει κάποια έρευνα σε σχέση με το τι έκανε η Ούνικ, η αποστολή του ΟΗΕ στο Κοσφοπέδιο και το εάν κάνει το ίδιο και η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η EULEX. Βλέπουμε πως στην EULEX υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ του προσωπικού γιατί υπάρχουν αφενός ε, υπάλληλοι και αφετέρου δίκαστες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εναλλαγή του προσωπικού, κάτι το οποίο βεβαίως δεν ωφελεί πάντα την εύρυθμη λειτουργία γιατί βεβαίως η Γιουλέξη είναι και η μεγαλύτερη αποστολή μας νομίζω στον τομέα της εξωτερικής ε, πολιτικής ε, και είναι όπως είπα πάρα πολύ μεγάλη η εναλλαγή του προσωπικού και δεν ξέρω εάν είναι καλό αυτό και τον Οκτώβριο δηλαδή τώρα θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η αποστολή ή όχι το τα βασικά προβλήματα βέβαια στο κοσμοπέδιο παραμένουν είναι όλο το σύστημα το δικαστικό, η καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, οι δυσκολίες που υπάρχουν στα δημόσια έργα, τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας που δεν έχουν ε, ξεκαθαρίσει. Συζητήσαμε λοιπόν και με τον κύριο Κούτσι, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ε, νομίζω πως μας έκανε μια καλή εντύπωση. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση επίσης με μέλη της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού του ε, Κοινοβουλίου του Κοσφοπεδίου και αυτού του οποίου θα λέγαμε Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη σχέση τους με το ελεγκτικό συνέδριο ή το αντίστοιχο όργανο, εν περιπτώσει, για να δούμε ποιες στάσεις μπορεί να γίνουν για να ενισχυθεί το έργο τους και ε, πλην ε, βεβαίως ε, της Πριστίνας πήγαμε και στο βορρά, στη Βόρεια Μητροβίτσα βεβαίως είναι δύσκολη η κατάσταση. Υπάρχουν τάραχες και δυσκολίες, αλλά βεβαίως ε, είδαμε όχι μόνο το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του κέντρου πληροφορίας, αλλά εκεί πέρα όπου πραγματικά έχει χτίσει σπίτια για τους ε, Ρώμα, τους Τσιγκάνους, οι οποίοι παλαιότερα ε, ζούσαν σε απαράδεκτες συνθήκες από πλευρά υγιεινής και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε νομίζω ολόκληρη αντιπροσωπεία από το τι γίνεται εκεί πέρα. Είδαμε και κάποια άλλα μικρότερα έργα όπου νομίζω πως το θετικό εκεί πέρα ήταν πως εντάξει είναι μικρά έργα αυτά δεν θα έχουν μεγάλη ε, επίπτωση, αλλά βεβαίως ε, για τους ανθρώπους τους οποίους ε, αφορούν θα είναι μεγάλη η αλλαγή στην ζωή τους για την επαγγελματική τους κατάρτιση ας πούμε, για να μπορέσουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Νομίζω πως είναι πολύ θετικά αυτά τα οποία είδαμε εκεί πέρα. Επίσης στην ΦΥΡΟΜ είδαμε την ε, κατασκευή ενός ε, αστυνομικού τμήματος στον, στο Τέτοβο που είναι πολυεθνική η κοινότητα και υπήρχαν ε, κάποιες εντάσεις αλλά τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες και είναι ένα υποδειγματικό έργο και χρηματοδοτείται από την προενταξιακή βοήθεια και ένα άλλο έργο επίσης γυναικών ε, για να καταπολεμηθεί το... η σωματεμπορία. Και οι κυρίες εκεί πέρα τις οποίες ε, στηρίζουμε νομίζω το εκτιμούν ε, πάρα πολύ. Και είχαμε και μια ενημέρωση με τον πρέσβη τον Πέτερ Σέρνσεν, τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας στα Σκόπια και τον άμεσο συνεργάτη του, όπου είδαμε στην πράξη πως ε, πράγματι υπάρχει αρκετός ε, συντονισμός, ε, αλλά βλέπουμε και τις δυσκολίες. Δημιουργείται ένας αυτοκινητόδρομος και πρέπει να υπάρχει συντονισμός με τις αρχές, με τις τοπικές αρχές επίσης, όπου υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Οπότε έχω καταλήξει από όλες μας αυτές τις εμπειρίες σε 23 συστάσεις και ελπίζω να τις ε, διαβάσετε και να τις δεχτείτε όλες. Νομίζω πως ε, θα πρέπει να το δούμε και στην επόμενη διαδικασία και να συμπληρωθεί την επόμενη φορά η αντιπροσωπεία και με συναδέλφους από το ΕΛΚ και τους φιλελευθέρους και ίσως θα μπορούσαμε μετά να κάνουμε ε, να απευθύνουμε γραπτές ερωτήσεις στην Κομισιόν ε, ή να έχουμε μια γραπτή επικοινωνία με την EULEX. Ε, αλλά βεβαίως αυτά καλά είναι, αλλά καλό είναι να πηγαίνουμε και επί τόπου να βλέπουμε το τι το τι γίνεται, γιατί βεβαίως ο εισηγητής ο οποίος ασχοληθεί με την απαλλαγή, νομίζω του χρόνου θα μπορέσει να επωφεληθεί από αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος από τους συναδέλφους που ταξίδεψαν μαζί μας, ο κύριος Σταυρακάκης ή κάποιος άλλος θέλει να συμπληρώσει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, αναμένω τις σα. Κύριε Σταυρακάκη. Thank you, Mr. President. You have presented the... Παρουσιάσατε την έκθεση με πάρα πολύ ολοκληρωμένο τρόπο και δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Eh, Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Η Κομισιόν διάβασε την ε, έκθεσή μας. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις. Ε. Όχι, μόνο βλέπω χαμόγελα. Ούτως ή άλλως ε, να σας πω πως η συνεργασία με την Κομισιόν Επιτόπου ήταν εξαιρετική και επί της όσον αφορά βεβαίως τις διατυπώσεις. Εντάξει, χαρούμενα. Χαρούμενα πρόσωπα. Ε, αν θέλετε, ευχαρίστω. Yeah. Ε, ε, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας στο Πέδιο και της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης επιβεβαιώνουμε αυτό που είπατε ότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με σας και την αντιπροσωπεία που επισκέφτηκε το Πέδιο και η ομάδα της Επιτροπής που ασχολείται εδώ και οι σύνδεσμοί μας επιτόπου μπορέσαμε να συζητήσουμε τα θέματα και με τη δική σας γραμματεία και τα σχόλια που είχαμε κάνει τα περισσότερα έλειφθαν υπόψη σε αυτά τα οποία λέτε. Γενικά είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Ωραία. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις τελειώνουμε και με αυτό το θέμα και φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασης αλλά βεβαίως οι συντονιστές ε, θα συνεχίσουν. Ε, προβλέπονταν για τις 6 ώρα, αλλά δεν ξέρω εάν οι επικεφαλής των ε, πολιτικών ομάδων μπορούν να δεχτούν να ξεκινήσουμε νωρίτερα, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Να κάνουμε 5 λεπτάκια λοιπόν διάλειμμα και ξεκινάμε και μισή με τους συντονιστές. 5, 5 και μισή λοιπόν.